Ah. Good morning, everybody. Looks like the Paris and and uh, Tuesday morning complicated our attendance, but. Καλημέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Η ώρα έχει περάσει, πρέπει να αρχίσουμε. Πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Υπάρχει μια μικρή τροποποίηση στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης. Πρέπει να συστήσουμε συζητήσουμε και τις συστάσεις των συντονιστών της 16ης Νοεμβρίου. Υπάρχει κάτι άλλο, κάποια αλλαγή, κάποια αντίρρηση. Ωραία, συνεπώς με την τροποποίηση αυτή εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Περνάμε στο δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που είναι οι ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Πρώτη μου ανακοίνωση να σας ενημερώσουμε για την αποστολή της ΕΝΒΙ στην 27η συνάντηση των ε, μερών, το ΜΟΠ 27, στο πρωτόκολλο του Μότρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν το στρώμα όζοντος. Επίσης στο Ντουμπάι, 3 με 5 Νοεμβρίου για τις επόμενες συνεδριάσεις μας. Θα έχουμε μια έκτακτη συνεδρίαση κοινή με την Άγκρη και την ΤΕΒΕ στη, την 5η 3 Δεκεμβρίου, 9.30 με 11.30. Εκεί θα ανταλλάξουμε απόψεις με τον ΦΑΟ, επί τη ευκαιρία του Διεθνούς Έτους για το έδαφος. Επίσης, έκτακτη συνεδρίαση της ΕΝΒΗ θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ελπίζω τουλάχιστον κατά τις 7 για να ψηφίσουμε τις ενστάσεις όσον αφορά τα μέτρα επιτροπολογίας για τις πραγματικές εκπομπές οδήγησης. Όσον αφορά την διερμηνία έχουν περισσότερες γλώσσες από ό,τι χρειαζόμαστε, από ό,τι φαίνεται, σε 22 γλώσσες. Όχι στα εστονικά, ούτε στα αγγέλικα όμως. Και βέβαια για όσους δεν είναι παρόντες στην αίθουσα, υπάρχει η αναμετάδοση μέσω διαδικτύου. Webstream. Επόμενο θέμα, σημείο 3 στην ημερήσια διάταξη. Εδώ πρόκειται για τις συστάσεις των συντονιστών έχουν κυκλοφορήσει ηλεκτρονικά. Σας έχουν σταλεί δηλαδή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρούνται εγκεκριμένε. Καλώ. Σημείο 4 στην ημερήσια διάταξη. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων της 3 η Σεπτεμβρίου 2015 και της 15 η Σεπτεμβρίου 2015. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει μέχρι το τέλο τη συνεδρίασή μα, τότε θα θεωρηθούν εγκεκριμένα. Επόμενο θέμα. Υποβολή έκθεση σχετικά με τις τρέχουσες διοργανικές διαπραγματεύσεις για διάφορα θέματα. Πρώτον, ιατροτεχνολογικά προϊόντα και διαγνωστικά in vitro ιατροχνολογικά προϊόντα. Βίλμοντ και Λίζε. Μετά τις διοργανικές διαπραγματεύσεις έγιναν δύο τριμερείς διάλογοι. 10 Νοεμβρίου του 2015 ήταν ο τελευταίος και η συμφωνία επί την αρχή επιτεύχθη όσον αφορά τους ορισμούς των διαγνωστικών αυτών μεθόδων. Επίσης προσωρινά μέτρα εγκρίθηκαν για να διακριθούν οι διάφορες περιπτώσεις βάσει του άρθρου 49. Ο τέταρτος τριμερή διάλογος έγινε τέλη Νοεμβρίου. Συζητήθηκαν τα θέματα τα οποία είχαν συζητήσει στους προηγούμενους τριμερείς διαλόγους. Η Προεδρία δεν μπόρεσε να στείλει συμβιβαστικές ε, προτάσεις 18 Νοεμβρίου έγινε ο τέταρτο τριμερή διάλογος. Τα θέματα τα οποία ε, συμφωνήθηκαν ήταν για τα μηχανήματα αισθητικής, για τις ε, εξαιρεσει και τους ορισμούς όσον αφορά τα Ιδρύματα Υγείας και την ηλεκτρονική καταχώρηση του UDI. Ο πέμπτος τριμερής διάλογος θα λάβει χώρα στις 3 Δεκεμβρίου. Το επόμενο θέμα είναι το εκπομπών και έγκριση τύπου για κινητήρες εσωτερικής καύσης που προορίζονται για μη οδικά κινητά μηχανήματα. Με τον τρίτο τριμερή διάλογο που έγινε στις 16 Νοεμβρίου, όλα τα βασικά θέματα του φακέλου συζητήθηκαν από τους συνομοδότες. Αποφασίστηκαν κάποια ζητήματα ε, που είχαν να κάνουν με τον, τους πρώτους δύο τριμερείς ε, διαλόγους όσον αφορά την εμπορία των μηχανημάτων και ειδικέ ε, προδιαγραφές και για τη δυνατότητα ε, αντικατάστασης μηχανών για το NRMM. Ο επόμενος τριμής διάλογος θα είναι 3 Δεκεμβρίου για τα επόμενα ανοιχτά θέματα που παραμένουν και για τα, τις εσωτερικές πλωτές μετακινήσεις και για το retrofitting. Το επόμενο θέμα είναι η μείωση των εκπομπών ρήπων από δικά οχήματα. Στο δεύτερο τριμερή διάλογο συζητήσαμε για τη μείωση των εκπομπών ε, βάσει της συνένεσης και προσαρμογής στη συνθήκη της Λισαβόνας. Επιβεβαιώθηκαν διάφορα ζητήματα και οι συζητήσεις όσον αφορά την προσαρμογή για την συνθήκη της Λισαβόνας τέθηκαν τάπητος και θα συζητηθούν παρετέρω τεχνολογικές λύσεις στον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων. Τέλος, έλεγχοι και άλλες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση εφαρμογή νομοθεσία για τα τρόφιμα και τι ζωοτροφέ και τον κανόνα για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, την υγεία των φυτών, το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό και τα φωτοπροστατευτικά προϊόντα. Ο πρώτο τριμερή διάλογο έγινε σε 9 Νοεμβρίου και έδωσε την ευκαιρία στους συνομοθέτες να συζητήσουν τα θέματα για τα οποία ήδη είχαν κάποιες συγκλίνουσες απόψεις και να αποφασίσουν για την μέθοδο εργασία και το χρονοδιάγραμμα. Τρεις τεχνικές ε, συναντήσεις επέτρεψαν ε, στις ε, διάφορες πλευρές να συζητήσουν και καθαρά τεχνικά ζητήματα. Ένας δεύτερος τεμερής διάλογος θα λάβει χώρα σήμερα το βράδυ. Λοιπόν, τώρα, ξαφνικά πρέπει να δώσω το λόγο στον εαυτό μου. Γιατί το επόμενο θέμα, το σημείο 6 στην ημερήσια διάταξη, είναι η ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106 του κανονισμού για τον κατάλογο χωροκατακτητικών ξένων ειδών. Όπως θα θυμόσαστε, ο σχετικός κανονισμός κατατέθηκε από την Επιτροπή στα τέλη του 2013. Και στη συνέχεια είχαμε πρώτη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο την Άνοιξη που, του 2014 που ήταν βέβαια και έτος εκλογών. Οπότε ήταν δύσκολο να έχουμε διαπραγματεύσει και να εγκρίνουμε τον φάκελο για το θέμα αυτό. Η πρόταση λοιπόν, έχει τον κατάλογο χωροκατακτητικών ξένων ειδών. Αυτή ήταν η καινοτομία και ήταν δύσκολο να διαπραγματευτούμε προηγουμένως χωρίς αυτό τον κατάλογο. Βέβαια, η κατάσταση τώρα είναι κάπως παράδοξη σήμερα. Και οι χώρες μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνήθηκαν να δεχτούν κατεξοδότηση πράξης για να καταρτιστεί ο κατάλογος αυτός χωροκατακτητικών ξένων ειδών. Τελικά επετεύχθη κάποια συμφωνία αφού σε τριμερή διάλογο αποφασίστηκε η κατεξοδότηση πράξη για το αξιολόγηση κινδύνου όσον αφορά τα είδη αυτά θα εγκριθεί πριν συνταχθεί ο κατάλογος. Κάτι το οποίο δεν έγινε. Και γι' αυτό υπάρχει ένσταση τώρα όσον αφορά τον κατάλογο αυτό. Οι λόγοι περιγράφονται στο κείμενο της ένστασης λεπτομερώς. Σήμερα δύο θέματα θα θίξω. Το ένα είναι η πρόταση για την καταξιότητα της πράξης όσον αφορά την αξιολόγηση κινδύνου. Και το δεύτερο είναι το αποτέλεσμα ενδεχομένως της προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις όσον αφορά την αξιολόγηση κινδύνου πρώτα. Η Επιτροπή έχει στείλει κάτι αφού κατατέθη η ένσταση, ένα πληροφοριακό σημείωμα δηλαδή, το οποίο λέει προκειμένου να λάβουμε υπόψη μας στις πρόσφατες εξελίξεις, ο κανονισμός προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει σε καταξιδότηση πράξη βάσει του άρθρου 5 σημείου για να διευκρινίσει παρετέρω τα στοιχεία εκείνα τα οποία επιτρέπουν να αξιολογήσουμε τα είδη εκείνα τα οποία μπορούν να οδηγηθούν σε χωρακακτικά ξένα είδη και να δώσει συγκεκριμένη περιγραφή των επιπτώσεων που πρέπει να ληφθούν υπόψη, προκειμένου να γίνει εξολόγηση κινδύνου. Κλείνω την παράθεση από το κείμενο της Επιτροπής. Φαίνεται σαν η Καταξιδότηση πράξη βάσει του 5.3 είναι κάτι που γίνεται σε θελοντική βάση, συμπληρωματικά, που διευκρινίζει κάποια μόνο στοιχεία. Και πάλι παραθέτω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μπορεί να χειριστεί σε ένα παρετέρω στάδιο. Βάσει του 5.3 αξιολόγηση είναι ζωτική σημασία για να υπάρξει διαφάνεια και συγκρίσιμη αξιολόγηση από πλευρά των χωρών νομελών... και άρα πρέπει να αναφέρονται όλα τα είδη τα οποία καλύπτουν τα πέντε κριτήρια που αναφέρονται στο 4.2. Η πρόθεση είναι, και εδώ ο κανονισμός λέει, κάτι που επίτηδες διπλωματικά παρέβλεψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λέει λοιπόν ο κανονισμός ότι πρέπει να δίνει λεπτομερή περιγραφή των επιπτώσεων τα σημείων α έως h της παραγράφου 1 και ότι η λεπτομερής περιγραφή θα αναφέρει και τη μεθοδολογία που πρέπει να χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη εθνικές και διεθνείς προδιαγραφές, αλλά και την ανάγκη κατά προτερότητα δράσεων για να αντιμετωπιστεί το θέμα των ειδών αυτών, τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν σημαντικό πρόβλημα στην βιοπικιλότητα ή σε άλλου είδους θέματα που έχουν να κάνουν με τα οικοσυστήματα. Οι διαπραγματευτές συμφώνησαν για εφαρμοστική πράξη και η κατεξιοδότηση πράξη είναι αναγκαία για να καθοριστεί ο κατάλογος των χωροκρατικών ξένων ειδών. Είναι εξοργιστικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρχεται και να λέει τώρα και παραθέτω ότι ο κανονισμός δεν αναφέρει και το λέω κατά λέξη γιατί από το σημείο 5.3 που σας ανέφερα πριν είναι σαφές ότι είναι αναγκαίο. Είναι επίσης σαφές ότι χρησιμοποιώντας ε, τέτοιες ασαφείς διαδικασίες καταλήγουμε και σε ασαφή αποτελέσματα. Χρόνια προσπαθούμε να καθορίσουμε τον κατάλογο των χωροκατακτητικών ξένων ειδών και θέλουμε να προχωρήσουμε. Οι καθυστερήσεις κοστίζουν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει και το σημείο 4-6. Τα αποτελέσματα πάντως είναι αδύναμα για μένα και το ξέρουν όσοι συμμετείχαν στη σύνταξη του καταλόγου που δεν είναι ικανοποιημένοι με τόσα περιλαμβάνει. Είναι ένας κατάλογος λοιπόν που κανένα χερσαίο είδος του DC100 δεν αναφέρεται. Ο κατάλογος αυτός δεν αναφέρει πολλά είδη. Το American Mink για παράδειγμα που είναι ένα από τα χειρότερα χωροκαθετικά ξένα είδη δεν αναφέρεται. ή κάποια άλλα από την Νότια Αμερική που ζουν ε, αλλού μακριά σε κάτι νησιά και δεν, και δεν υπάρχουν καν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρονται. Και δεν αναφέρονται άλλα τα οποία είναι πολύ πιο επικίνδυνα. Υπάρχουν και άλλα είδη που αναφέρει ο μιλητής, χωρίς όμως να τα αποκρίνονται στις προδιαγραφές. Ο μιλητή αναφέρει διάφορα είδη, τα οποία αναφέρονται και άλλα που δεν αναφέρονται. Όλη η εξολόγηση κινδύνου που γίνεται απορρέει μόνο από πολύ περιορισμένες πηγές. Γιατί είναι πρόβλημα τη στιγμή που ο κατάλογο μπορεί να συμπληρωθεί αργότερα. Η απάντηση είναι εξή. Έχω δουλέψει πάνω στα χωροκαθητικά ξένα ήδη πάνω από 20 χρόνια και μετά από την εμπειρία μου αυτή μπορώ να σας πω ένα πράγμα με βεβαιότητα. Για να υπάρχει εμπιστοσύνη και συνεργασία με το κοινό, μάλλον η εμπιστοσύνη του κοινού είναι προϋπόθεση για να πετύχει ο σκοπός μας. Ένα στραβό βήμα, μία κακή πρόταση πλήττει την εξοπιστία αυτή και την συνεργασία με το κοινό και χρειάζονται χρόνια για να ανακτηθεί αυτή η εμπιστοσύνη. Κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει λοιπόν στο κόσμο γιατί αναφέρονται κάποια φυτά του σημερινού για παράδειγμα και δεν αναφέρονται άλλα τα οποία καταστρέφουν τις δικές τους τις ε, καλλιέργειες. Η Επιτροπή είπε ότι δεν υπήρχε αρκετός χρόνος και περίμενα την κατεξοδότηση πράξη και έτσι υπονομεύτηκε το αποτέλεσμα του στόχου. Ναι, αλλά ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία υπέβαλε την ε, πρόταση με καθυστέρηση. Και πάλι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τον κατάλογο, ο οποίος μας αναγκάζει και εμάς να καθυστερήσουμε την διαδικασία και να πάμε βασικά πίσω χρόνια επειδή ακριβώ χάνεται έτσι η εμπιστοσύνη του κοινού. Συνεπώς Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πάτε πίσω την πρόταση αυτή, φροντίστε να υπάρχουν σωστέ προποθέσει για την αξιολόγηση κινδύνου και λάβετε υπόψη όλος όλο πρέπει να λάβετε υπόψη, εξηγήστε στις χώρε μέλη ότι υπάρχει και κόστος λόγω αδράνειας και ελάτε πίσω με μια καλύτερη πρόταση. Αυτά. Από το ΕΛΚ τώρα. Δεν βλέπω να είναι εδώ η συνάδελφος. Συνεπώς. Ποιος θα πάρει το λόγο. Μήπως μπορώ να πω κάτι διαδικαστικό, δηλαδή μήπως θα έπρεπε να ζητήσουμε από την Κομισιόν πρώτα να τοποθετηθεί εκείνη γιατί βεβαίως ε, μπορούμε όλοι να λέμε τα ίδια και τα ίδια αλλά ίσως θα ήταν καλύτερα πρώτα απ' όλα να ακούσουμε την Επιτροπή πριν τοποθετηθούμε εμείς. Πρόεδρος, νομίζω ότι αν δεν έχει ζητήσει κανείς άλλος ε, το λόγο και από ό,τι φαίνεται αυτό ισχύει. Ε, καλύτερα λοιπόν πράγματι να δώσουμε το λόγο στην Επιτροπή και μετά βλέπουμε. Βεβαίω αν συμφωνεί η Επιτροπή. Παρακαλώ, συμφωνείτε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ε, ευχαριστήσω που μας δίνετε τη δυνατότητα να εξηγήσουμε τη διαδικασία την οποία έχουμε εγκρίνει ε, προετοιμάζοντας ε, αυτό τον ε, κατάλογο των χωροκατακτητικών ειδών. Θα ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσω ότι η Κομισιόν είναι δεσμευμένη, απόλυτα δεσμευμένη, να εφαρμόσει τον σχετικό κανονισμό εκεί που γίνεται λόγος για τα χωροκατακτητικά είδη. Είπαμε λοιπόν στην ενδιάμεση έκθεσή μας για την στρατηγική βιοπικιλότητας ότι αυτός ο κανονισμός είναι καθοριστική σημασίας για να επιτύχουμε το στόχο μας μέχρι το 2020. Τώρα, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα που είναι να εγκριθεί αυτός ο κατάλογος το συντομότερο δυνατόν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η Επιτροπή των Περιφερειών έχουν τοποθετηθεί στην ενδιάμεση έκθεση, στην έκθεση Επιτροπής και εκεί αναφέρεται η έκκληση να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε αυτός ο πρώτος κατάλογος να εγκριθεί το συντομότερο δυνατόν. Διότι με τον τρόπο αυτό θα δραστηριοποιηθούν πολλά στοιχεία στην έκθεση και είναι σημαντικά αυτά. Καθίσταται απαραίτητο για τα κράτη-μέλη να θέσουν σε ισχύ τα απαραίτητα εργαλεία έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν τα σημαντικότερα στοιχεία του κανονισμού, παραδείγματο χάρη μέτρα αναχέτησης, μέτρα εγκύρη εκρίζωσης, ε, απαγόρευσης κ.ο.κ. Δεν θα ήθελα να αναφέρω όλα τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στο σημείωμα της Επιτροπής, αλλά θα μου επιτρέψετε να τοποθετηθώ κυρίως ορισμένα από αυτά που ελέγχθησαν. Παραδείγματο χάρη, να αναφερθώ λιγάκι την έγκριση του κανονισμού στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου. Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση να δοθεί εξουσιοδότηση στην Επιτροπή να εφαρμόσει κατεξουσιοδότηση πράξεις που θα διευκρινίζουν περαιτέρω ε, τα συγκεκριμένα μέτρα, αυτή η πρόταση προέρχεται προέρχεται κατ' ουσίαν από την Επιτροπή. Άρα δηλαδή δεν προέκυψε στο πλαίσιο του τριμερού διαλόγου, είχε γίνει από την Επιτροπή. Και η Επιτροπή πιστεύει ότι είναι σημαντικό να υπάρχει αυτή η εξουσιοδότηση. Και μάλιστα δεσμευτήκαμε να εφαρμόσουμε τέτοιε κατεξουσιοδότηση πράξει. Πρώτα απ' όλα όμω επιθυμούσαμε να ενημερωθούμε για τη διαδικασία σύσταση του καταλόγου. Δηλαδή ποια είναι τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν και με βάση το άρθρο 3, ποια είναι από αυτά που χρήζουν περαιτέρω διευκρίνηση το άρθρο 4.3 ε, συντάξαμε μία μελέτη όπου αναφέρουμε τι ακριβώς ε, σημαίνουν αυτά τα κριτήρια. Όλα αυτά τα συζητήσαμε με τους εμπειρογνώμονες και με την καθήλια αρμόδια επιτροπή. Επίσης, δεν συμφωνώ για το ότι η Επιτροπή δήθεν ε, συνέταξε τον κατάλογο μετά από πολιτική πίεση. Όχι. Εμείς ακολουθήσαμε αυστηρά τα κριτήρια τα οποία αναφέρει ο ίδιος ο κανονισμός ε, καθορίζοντας ποια είδη να συμπεριληφθούν στον κατάλογο και ποια όχι. Ένα λοιπόν από τα σημαντικότερα κριτήρια είναι ότι προβλέπεται μία αξιολόγηση κινδύνου ε, που ε, καλύπτει τα κριτήρια του 4-3, άρα δηλαδή υπάρχουν ε, πολλά είδη που αναφέρθηκαν, το American Mean, το Kundo, όπου πρέπει να σας πω ότι εκεί δεν ε, υπάρχει αξιολόγηση κινδύνου που να καλύπτει τα απαραίτητα κριτήρια. Και γνωρίζουμε μάλιστα ότι τα κράτη-μέλη εργάζονται επί του να βελτιώσουν περαιτέρω την αξιολόγηση κινδύνου. Και μόλις υπάρχει αξιολόγηση κινδύνου που θα καλύπτει αυτά τα κριτήρια, τότε η Κομισιόν προφανώς και δεν θα διστάσει να τοποθετήσει και αυτά τα είδη στον κατάλογο. Έτσι ώστε μετά ο κατάλογος να υποβληθεί στην καθήλυν αρμόδια επιτροπή. Υπάρχουν πολλά χωροκατακτητικά είδη που περιλαμβάνονται στο κατάλογο γιατί εκεί πράγματι έχει γίνει ε, αξιολόγηση κινδύνου. Water hyacinth. Αυτό ο είδο ε, προκαλεί τεράστιε ζημιέ ε, στον ποταμό Γουαρδιάνα και είναι πολύ σημαντικό να μην καθυστερήσουμε την έγκριση του πρώτου καταλόγου σχετικά ε, με τον Ιδροκιάκινθο που περιλαμβάνεται έτσι ώστε να μπορέσουμε να αναχαιτήσουμε την περαιτέρω επέκταση αυτού του ιδιαίτερα χωροπεκτητικού είδους του Ιδροϊάκινθου. Και υπάρχουν και άλλα που είναι ιδιαίτερα χωροκατακτητικά και αποτελούν μεγάλη απειλή για τη βιοπικιλότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν σκεφτήκαμε ότι δεν θα ήταν σκόπιμο πρώτα να προηγηθεί μια συζήτηση για τα κριτήρια, μα αυτά είναι ήδη σαφή στο κανονισμό, σκεφτήκαμε ότι είναι καλύτερα να ιδιαρχήσουμε τη δουλειά μας. Δηλαδή να καταλήξουμε στα είδη ε, που υπάρχει αξιολόγηση κινδύνου, να τα βάλουμε αυτά στον κατάλογο και μετά να εκδοθεί ταχύτατα ο κατάλογος. Έχουμε δεσμευτεί του χρόνου να επικαιροποιήσουμε τον κατάλογο όταν ε, πολλά από τα είδη που ανέφερε ο αξιότιμος πρόεδρος θα συνοδεύονται από αξιολόγηση κινδύνου που θα καλύπτει τα κριτήρια. Επίσης πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό να γίνει το συντομότερο δυνατόν. Τώρα, και ένα άλλο σχόλιο που αναφέρεται στο σχέδιο του ψηφίσματος ότι δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες ε, για το Κοινοβούλιο και για το ευρύτερο κοινό ε, σχετικά με την ακολουθούμενη διαδικασία. Εδώ θέλω να σε επισημάνω ότι όλα τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Επιτροπών, όλες οι μελέτες της Επιτροπής, μα και όλες οι σημαντικές πληροφορίες έχουν περάσει ε, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκεί που αναφέρεται η Επιτροπολογία, και επίση και στο μητρό της ίδιας της ε, Επιτροπής. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι έχουμε κοινοποιήσει όλες τις σημαντικές πληροφορίες στο κοινό και βεβαίως είμαστε και στη διάθεσή σας για να σας ε, δώσουμε πληροφορίες και θα συνεχίσουμε αυτό να το πράττουμε ε, θα δίνουμε τις απαραίτητες πληροφορίες στους ευρωβουλευτές. Εδώ θα ήθελα να σταματήσω, ανακεφαλαιώντας να πω ότι η Κομισιόν απαρέγκλητα ακολούθησε τον κανονισμό και ίσως υπάρχει ένα θέμα που πρέπει να επαναλάβουμε, ότι ο κανονισμός δεν αναφέρει ότι η κατεξουσιοδότηση πράξη η οποία διευκρινίζει τα στοιχεία Τη αξιολόγησης κινδύνου ότι αυτό είναι εκ των όνου κάνευ για την έγκριση του καταλόγου. Όχι, το ελέγξαμε αυτό με την νομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξέρετε, προβλέπεται μια καταληκτική ημερομηνία που έχει δοθεί στην Επιτροπή να υποβάλει τον κατάλογο και συγκεκριμένα μέχρι το αργότερο τη Δευτέρα Ιανουαρίου. Και ε, υπάρχει και άλλη μια ημερομηνία που αφορά τις κατεξουσιοδότηση πράξης, άρα δηλαδή δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για προαπαιτούμενο ότι πρέπει δηλαδή να εγκριθεί η κατεξουσιοδότηση πράξης πριν εγκριθούν τα κριτήρια και πριν ε, κατατεθεί ο πρώτος κατάλογος. Εμείς θεωρούμε ότι είναι πολύ καλύτερα τα κριτήρια αυτά να διευκρινιστούν περαιτέρω όταν θα έχουμε εμπειρία, όταν θα έχουμε εγκρίνει τον πρώτο κατάλογο που σας επαναλαμβάνω, περιλαμβάνει ήδη που συνοδεύονται από καλή αξιολόγηση κινδύνου με βάση τα κριτήρια που προβλέπει το άρθρο 4.3. Πολύ ωραία λέει ο πρόεδρος. Τώρα έχετε το λόγο. Τα μέλη της Επιτροπής έχουν το λόγο. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Είμαι η Ρενάτα Σόμερ σήμερα. Πρώτα απ' όλα, Έχω εδώ πέρα ένα σημείωμα, αλλά εντάξει δεν θα σας το διαβάσω. Νομίζω ότι όλοι ξέρετε ότι είναι ένα σημαντικό θέμα, ότι κοστίζει πολλά χρήματα κλπ. κλπ. Όμως, πρέπει να πω, όσον αφορά το κατάλογο, εκτός είπε η Επιτροπή, ότι εξακολουθώ να έχω αμφιβολίες για το κατά πόσο έχει οργανωθεί καλά το θέμα όσον αφορά την αξιολόγηση κινδύνου. Κυρίως κοιτώντα τα αποτελέσματα. Ακούω αυτά που μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λένε ότι δεν υπάρχουν πολλά είδη που έχουν καλύπτουν τις προϋποθέτες για την αξιολόγηση κινδύνου, όμως πολύ δύσκολα μπορεί κανείς να καταλάβει γιατί κάποια είδη δεν περιλαμβάνονται στο κατάλογο και κάποια άλλα υπάρχουν στο κατάλογο. Και έχω ένα σωρό παραδείγματα εδώ που δίνει η κυρία Σόμερα, αλλά θα σας δώσω τη δικιά μου εμπειρία. Αφήνω στην πάντα το σημείο σημείωμα και σας λέω τη δικιά μου εμπειρία. Τα ζώα που ζουν στο νερό Στη Σουηδία έχουμε τον ε, Αμερικανό αστακό, τον Αμερικάνικο αστακό, δεν αναφέρεται, το, του ειρηνικού τα μίδια, τα στρίδια, συγγνώμη, και διάφορα ψάρια. Τίποτα από όλα αυτά δεν υπάρχει. Ενώ για μας στη Σουηδία είναι πολύ σημαντικά. Από την άλλη μεριά υπάρχει το Fish, Μίλησα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άκουσα τι είπαν ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε δεν σημαίνει το ότι υπάρχει στον κατάλογο ένα είδος ότι πρέπει να σταματάμε να το έχουμε. Οπότε δεν καταλαβαίνω. Αν δεν έχει σημασία το αν είναι στον κατάλογο ή όχι, τότε τί; Τελικά δηλαδή αυτός ο κατάλογος δεν με καθησυχάζει. Αντίθετα, μου προκαλεί περισσότερες ανησυχίες για το που πάμε. Γνωρίζω ανθρώπους από τη δικιά μου εκλογική περιφέρεια που ανησυχούν. Και η μόνη αντίδραση όταν μιλάω για τον κατάλογο αυτό στη χώρα μου, είναι ανησυχία για είδη που υπάρχουν στον κατάλογο. Γιατί δεν τους βοηθά ο κατάλογος αυτός να αντιμετωπίσουν χωροκατακτητικά ξένα είδη που είναι πρόβλημα για αυτούς. Γιατί δεν υπάρχουν αυτά στον κατάλογο. Ωραία, δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε καλά ενημερωμένοι ή όχι, δεν θα το κρίνω αυτό, αλλά είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς τη λογική του καταλόγου αυτού μετά από μια διαδικασία που θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική. Οπότε εμείς στο ΕΛΚ δεν είμαστε πεπισμένοι έτσι όπως έχουν τα πράγματα τώρα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριος Γκεμπραντή. Από πού να ξεκινήσω. Από το θέμα της ε, στρατηγικής για την βιοποικιλία, επικοινότητα. Υπάρχουν κάποια κόκκινα φώτα, αλλά υπάρχουν και κάποια πράσινα. Όπως ε, αυτά μπορούν να μας βοηθήσουν στο να καταπολεμήσουμε τα χωροκατακτητικά αλλοχθονά είδη. Στα χαρτιά όλα φαίνεται ότι είναι εντάξει. Και περιμένουμε την επόμενη φάση λοιπόν προκειμένου να πραγματοποιηθούν αυτά που βρίσκονται στα χαρτιά σε ό,τι μας αφορά λοιπόν αυτό που πράττει τώρα η Κομισιόν είναι κάτι το οποίο εμείς αναθέσαμε δώσαμε εντολή και είναι αρκετά στενή η προθεσμία μέχρι τις 2 του Ιανουαρίου προκειμένου να συντάξει το πρώτο κατάλογο των χώρο κατακτηριτών αλόφθονων ειδών. Αυτός ο κατάλογος που το παρόν είναι τέλειος, όχι, κάθε άλλο. Ένα παράδειγμα, στην χώρα μου, στην Ολλανδία, υπάρχουν τεράστια προβλήματα με το red Το καταπολεμούμε εδώ και καιρό, όχι επειδή δεν μας αρέσει, αλλά διότι επηρεάζει Αλλά ήδη και τώρα στον κόπο που ξεκίνησε στο Παρίσι συζητούν διάφορα ευαίσθητα ζητήματα και το μάσκρατ ε, παίζει σημαντικό ρόλο διότι επηρεάζει Red is not on the list right now. Τα Λοιπόν, γι' αυτό έχω ένσταση για τον κατάλογο. Θα πρέπει να αποφύγουμε το ότι το καλύτερο είναι εχθρός του καλού. Η προδεσμή η οποία υπάρχει και τους έχουμε ζητήσει να έρθουν με ένα σχέδιο έκθεσης πριν από τις 2 Ιανουαρίου. Το κατάλογος λοιπόν δεν είναι τέλειος ε, κάθε άλλο, αλλά όπως είπε η Κομισιόν υπάρχουν επαρκή εργαλεία για να προσαρμοστεί ο κίνδυνος, ε, ο κατάλογος συγγνώμη, στο, τα επόμενα έτη. Ένα ζήτημα το οποίο Έφυξαν οι δύο συνάδελφοι οι οποίοι υπέβαλαν την ένταση. ανέφερε ότι βασίζεται σε πολιτικά κριτήρια και όχι σε επιστημονικά. Εγώ δεν είμαι επιστήμον, θα πρέπει λοιπόν να βασιστώ σε αυτά που λένε άλλοι. Αλλά γνωρίζω ότι εξετάσαμε τον κατάλογο ο οποίος ε, εξορισμού περιέχει και κάποια πολιτικά κριτήρια. Ο συνάδελφος Φιέλνερ είπε ότι μιλούσε όχι αποκλειστικά με βάση τον κατάλογο αλλά και με βάση την ε, εμπειρία του. Φαντάζομαι ότι και αυτό είναι μια πολιτική αξιολόγηση, πολιτική κρίση. με που έχουμε αυτή τη συζήτηση τώρα διότι έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην Κομισιόν και με εκπλήσει επίσης και ο συνασπισμός ο οποίος έχει δημιουργηθεί κατά αυτού του καταλόγου αισθάνομαι ότι άλλοι επιθυμούν έναν μακρύτερο κατάργο για άλλοι έναν πιο σύντομο ορισμένοι επιχειρηματολογούν λέγοντας ότι η Κομισιόν έκανε εξαίρετη δουλειά δεν θέλω να ασκήσω καμία κριτική και με διότι η ομάδα μου θέλει να δώσει την Κομισιόν τον ε, κάποια εύσημα για την προσπάθεια που κάνει για το ζήτημα του καταλόγου χωρακτακτικών ξένων ειδών να πω ότι η ομάδα μου, οι φιλελεύθεροι, θα καταψηφίσουν αυτή την ένσταση αν λάβουμε υπόψη τη βιοπικιλότητα στα σοβαρά και αν λάβουμε υπόψη την ε, αξιολόγηση της ε, λόγω στρατηγικής είμαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να ε, παρεμποδίσουμε αυτόν τον κατάλογο των χαρακτηριστικών όλων των ειδών και θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες ε, τα επόμενα χρόνια και να μην καταψηφίσουμε αυτό το σχέδιο καταλόγου. λόγο. Νομίζω λοιπόν ότι το χρονοδιάγραμμα για την Επιτροπή πράγματι ήταν πολύ φιλόδοξο και τα προβλήματα τα οποία αναφέρθηκαν σήμερα έχουν σχέση με αυτό το χρονοδιάγραμμα. Όσον αφορά τη σύνταξη του καταλόγου, μόνο το 1 τρίτο πετύχαμε και το βασικό πρόβλημα οφείλεται στο ότι εφαρμόστηκαν διαφορετικά κριτήρια, ως εκ τούτου το αποτέλεσμα είναι εμβαλωματικό, δεν καταδεικνύει συνέπεια. Δεν τα βρίσκω ικανοποιητικά αυτά που μας είπατε. Υπάρχουν λοιπόν τρία προβλήματα που κατά την άποψή μου είναι απόλυτα ξεκάθαρα. Καταρχάς, το ερώτημα ένα είδος πότε είναι χαρακτητικό, ε, πότε πρέπει να λάβουμε μέτρα. Ε, βεβαίως και αυτό είναι θέμα κόστους, η Κομισιόν το ανέφερε αυτό. Ε, πρέπει να δούμε λοιπόν ποιο είναι το κόστος που προκύπτει από αδράνεια. Η Κομισιόν όμως και αυτή δεν έχει πει αυτό που πρέπει, δεν έχει δώσει απαραίτητες πληροφορίες, άρα δεν μπορούμε να υπολογίσουμε το συνεπακόλουθο κόστος. Πιστεύω ότι ο ελάχιστος στόχος είναι το να μην επεκτατούν περαιτέρω χωροκατακτητικά είδη. αυτό είναι ο πρώτος στόχος. Και όχι τόσο η ε, καταπολέμηση χωροκτατητικών ειδών, γιατί αυτά υπάρχουν εδώ και πολύ καιρό. Με το να ε, αντιμετωπίσουμε περισσότερο την αναστολή θα έχουμε μεγαλύτερη επιτυχία. Αυτό ήταν το δεύτερο. Τώρα, το τρίτο είναι το εξής. Η σύνταξη του καταλόγου αφορά ε, ενιαία κριτήρια και όχι τα διάφορα που ακούστηκαν εδώ, που όπως σας είπα όλα αυτά μας οδηγούν στο να έχουμε μια εμβαλωματική εντύπωση. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, πιστεύουμε ότι δεν είναι σωστό να προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Από την άλλη πλευρά βέβαια πρέπει να πούμε ότι αναμφίβολα πρέπει να γίνει το πρώτο βήμα για να ακολουθήσουν ε, ταχύτατα και το δεύτερο και το τρίτο να προχωρήσουμε και τα κράτη-μέλη καλούνται ε, να υπολογίσουν όπως σας είπα το συνεπακόλουθο κόστος. Πολύ ωραία λέει ο Πρόεδρος. Η Ευχαριστώ πολύ ως ε, μέλος αυτής της ε, παράδοξης ε, συμμαχίας ήθελα και εγώ να πω ορισμένα πράγματα. Ζητώ συγγνώμη που ήρθα καθυστερημένη και δεν άκουσα τι είπε η Επιτροπή. Μετά βέβαια θα ενημερωθώ. Κοίταξε, εμένα αυτό που με απασχολεί κυρίως είναι το εξής, ότι βεβαίως και έχουμε αντιρρήσεις και επειδή ήμουνα σκιώτη εισηγήτρια από αυτού στην προηγούμενη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μιλήσαμε πάρα πολύ για το θέμα γιατί όταν είναι κανεί σκιώτης εισηγητής προφανώς και κάνει τον κόπο να ενημερωθεί ε, για προβλήματα ε, γενικά για τα είδη, τα ζώα, τα φυτά ε, ασχολείται κανείς με το τι γίνεται στο κράτος του αλλά και σε άλλα κράτη-μέλη. Τα έκανα λοιπόν όλα αυτά και έτσι αποκόμισε έτσι λίγο μια ιδέα ε, για το τι θα έπρεπε να περιμένω από αυτόν τον αρχικό κατάλογο. Και όταν ήρθε ο κατάλογος σοκαρίστηκα γιατί ανακάλυψα ότι κυρίως φυτά φυτά είναι εκείνα για τα οποία είχαμε συζητήσει και κάπως είχαμε καταλήξει ότι αυτά οπωσδήποτε θα εμφανιστούν στο κατάλογο και δεν εμφανίστηκαν. Καθαρά τεχνικά λοιπόν υπάρχουν λόγοι γιατί συνέβη αυτό αυτό ε, οφείλεται ίσως στην αξιολόγηση κινδύνου, αλλά εάν τελικά προκύπτει αυτός ο μη ικανοποιητικός κατάργος, που είναι κατά την απόψη μου μη ικανοποιητικός τώρα πρέπει να τον αλλάξουμε. Συμφωνώ με προαλήσαντες που είπαν ότι θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση στην Κομισιόν για να υποβάλει ένα καλύτερο κατάλογο. Σε αυτή λοιπόν τη συγκεκριμένη περίπτωση, περίπτωση ο τρόπος για να ασκήσουμε πίεση είναι να απορρίψουμε τον κατάλογο. Γιατί αν περάσει ο κατάλογος, αναγκαστικά ε, θα καθυστερήσει η διαδικασία. Πρέπει λοιπόν να στείλουμε ένα μήνυμα στα κρατημέλη ότι αυτό το θέμα πρέπει να το εξετάσουν πιο προσεκτικά. Ε, το θέμα δεν είναι να αποφύγουμε εκείνα τα είδη που κοστίζει πάρα πολύ για να τα ξεριζώσει κανείς. Ε, είμαι λοιπόν ευτυχής που θα καταψηφίσω. Ελπίζω να μην υπάρξουν πια καθυστερήσεις. Ε, πιστεύω ότι ε, πρέπει κανείς να το σκεφτεί περισσότερο το θέμα και να ε, λάβει περισσότερα μέτρα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στη ρίζα του. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν βλέπω να ζητάει κανείς άλλο το λόγο και ως εκ τούτου ίσως μπορώ να δώσω το λόγο και πάλι στην Επιτροπή, για λίγο βέβαια, ε, για να τοποθετηθεί η Επιτροπή, αν θέλει βέβαια. Η Επιτροπή. Νομίζω πως ε, όλοι συμφωνούμε ότι ο κατάλογος δεν είναι πλήρης. Να σας πω ότι υπάρχουν ακόμα κάποιοι που θεωρούν ότι υπάρχουν πολλά είδη, άλλοι που θεωρούν ότι είναι λίγα τα είδη που περιλαμβάνει ο κατάλογο. Θα πρέπει όμως να διασφαλίσουμε πως ε, τα κριτήρια τα οποία έχουμε θέσει πληρούν τις ε, απαιτήσει. Ο Αμερικανικός ε, αστακός γνωρίζουμε ότι προετοιμάζεται μια, μια αξιολόγηση κινδύνου, μια μελέτη κινδύνου Τώρα για το Grey Fish υπάρχει στον κατάλογο διότι υπάρχει πλήρη αξιολόγηση κινδύνου και υπάρχουν πολλά κοινωνικο-οικονομικά επιχειρήματα για να μην συμπεριληφθεί στον κατάλογο. Έχουμε συζητήσει περί αυτού. Πιστεύουμε όμως ότι αξίζει τον κόπο να συμπεριληφθεί διότι πρέπει να αποφύγουμε να μην επεκταθεί περαιτέρω και στην Σκανδιναβία τα κράτη-μέλη όπου ε, το ίδιο αυτά υπάρχουν, έχουν κάποια προγράμματα για να μην υπάρχει περαιτέρω ε, περαιτέρω επέκταση αυτών των ξένων ειδών και ειδικά δεν θα πρέπει να επεκταθούν σε περιοχές που ήδη δεν υφίστανται. Πρέπει να αποφύγουμε επίσης ε, να φτάσουν σε νησιά όπου θα κάνουν μεγάλη καταστροφή. Πιστεύουμε λοιπόν ότι ο κατάλογος ε, σε ό,τι φορά τις επιστημονικές γνώσεις που έχουμε είναι κατάλληλος. Θέλουμε να, να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας και τις προθεσμίες και είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε συμπεριλάβει ήδη ε, τα οποία ε, πληρούν τις προϋποθέσεις αλλά είμαστε πρόθυμοι να βελτιώσουμε περαιτέρω τον κατάλογο όταν έχουμε αξιολόγηση κινδύνου για περισσότερα Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που ακούω ότι η Κομισιόν ε, θέλει να ε, σεβαστεί τις προθεσμίες και θα έχουμε μια συνάντηση με τον Επίτροπο και θα του θέσουμε ερωτήσεις και για διάφορους άλλους φακέλους. Εάν ε, παραστεί ανάγκη να εφαρμοστούν οι κατεξότηση πράξης ε, αυτή η συζήτηση θα είναι παροχημένη. Αυτή η συζήτηση γίνεται διότι δεν υπάρχουν κατεξότηση πράξης για μέρη αξιολόγησης κινδύνου. Δεν ξέρω αν θα έχουμε έναν μικρότερο ή μακρύτερο κατάλογο. Εμείς θέλουμε έναν σωστό κατάλογο, έναν καλό κατάλογο. Κάποιος είπε ότι το καλύτερο είναι εχθρός του καλού. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά δεν έχουμε έναν καλό κατάλογο. Λάθος ε, κατάλογοι θα μας οδηγήσουν σε λάθος αποτελέσματα και έλλειψη εμπιστοσύνης από το κοινό. Είμαι πεπισμένος πως ε, είναι πολύ καλύτερο να έχουμε αργότερα έναν κατάλογο παρά να έχουμε σύντομα έναν καλό κατάλογο ένα κακό κατάλογο. Αυτή η άποψή μου λοιπόν θα ψηφίσουμε στο ζήτημα αυτό το απόγευμα μετά τις 4 και θα περάσει την Ολομέλεια στις, ε, στη δεύτερη Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Επόμενο θέμα στη μισή διάταξη όπου και πάλι πρόκειται για μια ένσταση που αφορά την έγκριση γενετικά τροπημένου ΝΙΚΑΠΑ ΝΚ603 ΤΑΦ 25 να δώσω το λόγο στους υποβάλλοντες στην έσταση ο Μπαρτ Τάιζ έχει το λόγο Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι μαζί με τον Κιγιώμο Μπαλά Μπόιλαν και την Λεωνόρα Εύη Έχουμε μια πρόταση κειμένου όσον αφορά την ένσταση για την εφαρμογή του Σχεδίου Εφαρμοστικής Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται λοιπόν για τον αραβόσιτο γενετικά τροποποιημένο NK603-XT25. Πρόκειται για το πρόβλημα του γλυφοσάτ και του γλυφοσυνικού αμμονίου. Υπάρχει από την ΕΦΣΑ, από την Ευρωπαϊκή δηλαδή, Υπηρεσία Ασφάλειας Τροφίμων, θετική γνωμοδότηση, ε, που απαγορεύει όμως την καλλιέργειά του. Έχουμε συζητήσει για την απόφαση της ε, οργάνωσης κατά του καρκίνου που σε δικές της μελέτες έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μπορεί να πρόκειται για καρκινογενή ουσίες. Καρκινογενείς ουσίες. Βέβαια είναι πολύ τεχνικό το ζήτημα, δεν θα μπω ε, στις λεπτομέρειες. Πάντως το πιο βασικό επιχείρημα είναι πολιτικό και αυτό θα χρησιμοποιήσω. Από την αρχή με την Επιτροπή Γιούνκερ, ο ίδιος ο κύριος Γιούνκερ στις 15 Ιουλίου είχε πει ότι δεσμεύεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην πάρει αποφάσεις και να μην επιτρέψει προϊόντα με τα οποία διαφωνούν οι περισσότερες χώρες. Το νομοθετικό πλαίσιο λοιπόν μέσα στο οποίο ε, λειτουργούμε σήμερα επιτρέπει γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Δεν λειτουργεί λοιπόν καλά το σύστημα, δεν υπάρχει πλειοψηφία στο Συμβούλιο υπέρ. Έχουμε κάνει και εδώ τη συζήτηση πριν από μερικούς μήνες για την πρόταση την νομοθετική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και στην Ολομέλεια έχουμε πει ότι δεν λειτουργεί το σύστημα και στην Ολομέλεια ζητήσαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθει με νέα πρόταση. Πιστεύω λοιπόν ότι αν εμείς στην Ολομέλεια με ισχυρή πλειοψηφία αποφανθούμε κατά, τότε η αδειοδότηση για νέους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς δεν θα προχωρήσει. Είναι σαφές ότι πρέπει να πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει και που τη ζητάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που το έχει υποσχεθεί ο πρόεδρος ο ίδιος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Γιούνκερ. Συνεπώς πρέπει όλοι μαζί να στηρίξουμε το κείμενο αυτό που και με την ΚΟΕ και με τους σοσιαλιστές και με το FTD συμφωνήσαμε να το στηρίξουμε όταν ψηφίσουμε στις 4 το απόγευμα εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Πρόκειται για μια κοινή συζήτηση, όμως έχουμε και μια άλλη ένσταση για το ίδιο θέμα, οπότε θα έπρεπε να δώσω το, το λόγο και στην ε, άλλη βουλευτή που επίσης έχει ένσταση, την κυρία Κοντίν. Ευχαριστώ, ε, ε, την κυρία, συγγνώμη, τον Άνω. Ε, μιλάω εκ μέρους της κυρίας Γκοντίν, λέει κυρία Άνο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να επιτρέψει την εισαγωγή στην ευρωπαϊκή αγορά προϊόντων που περιλαμβάνουν γενικά τροποποιημένα αραβόσιτο NK603 ε, αυτό το αραβόσιτο το παράγει η Μονσάντο και τροποποιήθηκε για να είναι αρθεκτικό στα φυτοφάρμακο σύμφωνα με, με τη ε, χρήση του γλυφοσάτ και το οποίο βρίσκεται στο Wundop ένα φυτοφάρμακο το οποίο χρησιμοποιείται ευρύτατα στον κόσμο. Το, η ουσία αυτή, η γλυφοσάτ, είναι ανησυχητική και μόνο ότι η νομοδότηση της ΕΦΣΑ είναι, είναι αφήσιμη διότι δεν αφορά ακριβώς το γλυφοσάτ ε, και τις αποτελέσματα που έχει ε, για τον ε, καρκινογόνο επιρροή, επίδραση που έχει στους οργανισμούς των ανθρώπων. Ο... Έχει θεωρηθεί ως πιθανό καρκινογόνο καρκινογόνος ουσίας και αφορά όχι μόνο την υγεία των γεωργών αλλά και την βιοπικιλότητα των εδαφών και τα ζώα που ή τους που βόσκουν στις περιοχές. Ο καθένας θα έχει τη γνώμη του όταν γίνει η ανταλλαγή με τον ΕΦΣΑ. Τα προϊόντα που περιέχουν γλυφοσάτ είναι επικίνδυνα για τον οργασμό και για τη φύση. Κάθε φορά που βαίνει στην αγορά ένα προϊόν που περιέχει γλυφοσάτ, αυτό ε, επιδεινώνει περαιτέρω την κατάσταση οι Αμερικανικές αρχές ε, είναι απόλυτες. Περνάμε από 426 γραμμάρια ανά εκτάριο σε 1318 ανά εκτάριο για τους ε, γενετικά τρομενούς οργανισμούς. Διερωτώμεθα σε ποιον ωφελεί αυτό το προϊόν, ποιο είναι το συμφέρον για τους Ευρωπαίους. Η γεωργία τους ε, θα επηρεαστεί η αξιολόγηση των του που περιέχει τροπημένου θα έχει αμφίσιμα και αφίβολα αποτελέσματα. Και εδώ υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα για την αξιολόγηση. Δεν πρόκειται για την εξουσιοδότηση ενός προϊόντος που είναι γενετικά τροποποιημένο θα πρέπει να αξιολογηθεί ως ε, τέτοιο είδος ε, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ε, γεωργία. Όταν πρόκειται για τη μέτρηση της ρήπανσης, οι μηχανές των οχημάτων θα πρέπει να γίνονται και ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται κάτω από πραγματικές συνθήκες γιατί να μην χρησιμοποιηθεί η ίδια τακτική και για τα ε, γενετικά προϊόντα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν βέλτιστες πρακτικές και ενάρετες για την εισαγωγή αυτών των προϊόντων. Η εισαγωγή ε, γενετικά τροποποιημένων ειδών ε, αναφέρεται στην έκθεση του, της ε, Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών και αποδίδει και αφορά τα ζυζανιοκτώνα, τα φυτοφάρμακα τα οποία είναι όλο και πιο επικίνδυνα, όλο και πιο ακριβά και με καταστροφικές συνέπειε. Η περίπτωση του γλυφοσάτ, το οποίο αναμειγνύεται με την ουσία 2K2 και αυτή αποτελεί η ένσταση που έχει παρουσιάσει ο συνάδελφος Πάβελ Πόκ. επίσης να σας αναφέρω ότι το προϊόν της εταιρεία DOF που και αυτό περιέχει γλυφοσάτ ε, ε, έχει αποσυρθεί από την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών ενώ έχει εξουσιοδοτηθεί την περασμένη χρονιά διότι καταστρέφει την ε, χλωρίδα Αυτές είναι οι επιπτώσεις των ε, γενετικά προβλημένων οργανισμών. Κάθε φορά λοιπόν που εισαγάγει η Ένωση ε, τέτοια προϊόντα από τρίτα κράτη μας δημιουργούν πρόβλημα αδειοδοτώντα την εισαγωγή των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών ε, οδηγούμε σε υποδούλωση τους ε, γεωργού μας. Έχουν υποβληθεί διάφορα ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί ακόμα, κάτι το οποίο σημαίνει ότι η απάντηση της ε, ΕΦΣΑ δεν μπορεί να δοθεί σίγουρα με την οδηγη 1829 του 2003 και ακόμα και η περιεκτικότητα σε γλυφοζάτ είναι επικίνδυνη. Πέραν ε, τούτου και σε αντίθεση με την αρχή της πρόληψης ε, η Κομισιόν θεώρησε ότι θα πρέπει να εγκρίνει ε, τα προϊόντα αυτά που περιέχουν γλυφοζάντο. θεωρώ ότι έχει υπερβεί τα σεξουσίες της και ως εκ τούτου ζητώ να μην αδειοδοτηθεί η εισαγωγή του NK 603 ΤΑΦ 25. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Για το θέμα της συζήτησης και για τους γενετικά τοπομένους οργανισμούς, ξέρουμε ότι δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ μας σήμερα ούτε μεταξύ των ομάδων, ούτε ακόμα και μέσα στην ίδια ομάδα πολλές φορές. Εγώ είμαι απόλυτος, αλλά δεν είναι αυτό που μας απασχολεί σήμερα. Το πραγματικό πρόβλημα είναι πολιτικό. Έχουμε συζητήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη θέλησή της να επανεθνικοποιήσει την αδειοδότηση διάθεση στην αγορά γενετικά τροπημένων προϊόντων. Ιτήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό σημαίνει ότι απορρίφθηκε η πρότασή τη Και όχι μόνο απορρίφθηκε, γιατί θυμίζω ότι ψηφίστηκε και μια τροπολογία που ζητούσε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο γίνεται πιο γρήγορα να έρθει με νέα πρόταση. Είμαστε νομοθετικό σώμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εκτελεστικό σώμα. Συνεπώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολιτικά πρέπει να λαμβάνει υπόψη αυτά που εμεί λέμε. Αλλιώ τι νόημα έχει η ύπαρξή μα. Πέρα από αυτό, υπενθυμίζουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν μπορεί να συνεχίσει business as usual, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα, να συνεχίζει να δίνει άδεια σε γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, αν προηγουμένως δεν επανακαθορίσει το νομοθετικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δρά. Συνεπώς, Περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθει σήμερα με πρόταση για το αναγκαίο πλαίσιο προκειμένου να λαμβάνονται αποφάσεις για τη διάθεση στην αγορά, για την αδειοδότηση δηλαδή γενετικά τροπημένων οργανισμών και στο μεταξύ ζητάμε τόσο σοβαρές αποφάσεις όπως είναι η διάθεση στην αγορά γενετικά τροπημένων οργανισμών όσες διαφωνίες και αν υπάρχουν μεταξύ μας να μην λαμβάνεται υπόψη. Πρέπει να το πω και να το επαναλάβω και οι σοσιαλδημοκράτες αυτό ακριβώς στηρίζουν. Επόμενος, ο μιλητής η κυρία Εύη. Συγγνώμη, άκουσα άδει. Θα είμαι πολύ σύντομη. για να αναφέρω την ε, στήριξή μας ε, ως ε, ομάδα των πέντε αστέρων για την κατάσταση που βρισκόμαστε σχετικά με την εξέταση αυτού του θέματος, σχετικά με την εξουσιοδότηση των, των οργανισμών. Θα πρέπει λοιπόν ε, να υποβάλουμε ενστάσεις και στις επόμενες, επόμενα αιτήματα διότι το ζήτημα αυτό είναι πολύ σημαντικό το οποίο θα πρέπει να διευκρινιστεί το συντομότερο γι' αυτό είναι ένα στενερό μήνυμα που το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Περιβάλλοντος θα πρέπει να στείλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν με σθένος στηρίζω τις ενστάσεις των συναδέλφων που μίλησαν πριν από μένα. Ευχαριστώ. Φίλνερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι πολύ λυπηρή η συζήτηση αυτή. Την είχαμε και στο παρελθόν και νομίζω ότι θα την έχουμε και στο μέλλον. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν εξαντλείται ποτέ. Όταν μιλάμε για τους γενετικά τροπημένους οργανισμούς, η ΕΦΣΑ ήταν σαφέστατη, δήλωσε ότι δεν υπάρχει υψηλή κίνδυνη σε σχέση με τον ναραβόσιτο. Το 2003 η ΕΦΣΑ είπε εντάξει για το πρώτο θέμα και δεύτερη φορά το 2009 δήλωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ε, μεγαλύτερος από ότι σε ένα φυσικό προϊόν μη τροποποιημένο. Και μετά επανέλαβε ότι όχι δεν υπάρχει κίνδυνος ε, και τον Ιούνιο φέτος ε, είπε ότι ο συνδυασμός αυτών των δύο προϊόντων για τα οποία μιλάμε τώρα είναι ε, εξίσου ακίνδυνος όπως και το φυσικό προϊόν. Το όταν άκουσα τη συζήτηση αυτή με κάνει να σκέφτομαι αυτούς που οποίοι αρνούνται πως υπάρχει αλλαγή του κλίματος. Ε, ζήσαμε σε επιστήμονες να κάνουν σχετική αξιολόγηση και ακόμα κι αν ε, για 5, 10, 15 χρόνια επαναλαμβάνουν τα ίδια πράγματα, ε, φτάνει κάποιο ο οποίο λέει: Μα έχω του δικού μου εμπειρογνώμονε, οι οποίοι μπορεί να μην είναι πολλοί, αλλά πιστεύουν και υποστηρίζουν το αντίθετο. Εγώ του έχω εμπιστοσύνη. Νομίζω λοιπόν ότι αυτός δεν είναι ο σωστός τρόπος για τη λειτουργία της Επιτροπής μας. Θα πρέπει να αποφασίσουμε για να βρούμε τους εμπειρογνώμονες, να τους ακούσουμε και να ακολουθήσουμε τις συστάσεις τους. Διαβάζοντας τα επιχειρήματα εδώ και άκουσα επίσης ότι θα πρέπει να το δούμε το θέμα και από πολιτική σκοπιάς. Νομίζω ότι το μόνο που απομένει είναι αυτό όντω. γιατί αφού έχουμε εξετάσει όλες, τα τεχνικά και επιστημονικά ζητήματα και διαβάζοντα τώρα την ουσία βλέπουμε ότι η πρόοδο ε, δεν είναι ικανοποιητική, δεν έχει υπάρξει ειδική πλειοψηφία από τα κράτη-μέλη για την έγκριση αυτή τη εισαγωγή ε, αυτών των ε, γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Και Ρωτώ με αν αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο μπορούμε να υποβάλουμε σε, οποιοδήποτε άλλη, σε μια οποιοδήποτε άλλη συζήτηση και άλλο πλαίσιο. Εντάξει, υπάρχουν κάποια κράτη τα οποία δεν συμφωνούν, αλλά γνωρίζουμε ότι ψηφίσαμε τι προτάσει της νέας κομισιόν, της η οποία ε, ε, για διάφορου λόγου. Αλλά αυτό να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα λέγοντας ότι καταψηφίσαμε την προηγούμενη, για αυτό λοιπόν θα πρέπει να σταματήσουμε οποιαδήποτε χρησιμοποίηση και εισαγωγή αυτών των ε, προϊόντων. Ε, το, το μορατόριο δεν ε, πέρασε, άρα θέλουμε να ε, βάλουμε τώρα το, ένα μορατόριο από την πίσω πόρτα. Αυτό είναι αντίθετο με αυτό όπω στην Ολομέλεια. Αν κοιτάξουμε λοιπόν το τι λένε οι επιστήμονες και οι υπερογνώμονες, εμείς αποφασίσαμε πάνω σε αυτά που μας είπαν. Ακόμα και αν ε, σε πολλούς δεν αρέσει αυτή η νομοθεσία, εμείς συμφωνήσαμε με την νομοθεσία. Ποτέ δεν ε, υπήρξαν τόσοι πολλοί πράσινοι υπουργοί στο Συμβούλιο. Α, όταν, παρά, όταν ε, εγκρίθηκε αυτή, αυτό το νομοθέτημα και τώρα δεν μπορούμε να το μπλοκάρουμε και να σταματήσουμε την όλη διαδικασία από την πίσω πόρτα. Θα πρέπει να πούμε λοιπόν ότι είναι ανεύθυνο να ε, κάνουμε το μορατόριο και να το συμπεριλάβουμε από την πίσω πόρτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Νίλ Στόραντ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, λοιπόν, να τα πούμε με μια κουβέντα. Χάλια. Χάλια όλα. Και καλύτερα να πάμε για καφέ. Η αντίρρηση της κυρίας Γκούντενς είναι κάτι ε, που εμείς ε, στα σουηδικά θα το λέγαμε έτσι σε ελεύθερη μετάφραση Τύρδιν μίγδιν, πλην φιλήθη κέραμια, ατάκτου ερημένη. Λοιπόν, κατανοώ ε, το μοραλιστικό στοιχείο, αλλά δεν κατανοώ τη διαδικασία. Όσον αφορά τις αντιρρήσεις μας, κοιτάξτε και εμείς ε, ηθικοπλαστικής και ηθικολογικής είναι η αντίρρησή μας. Εγώ προσπαθώντα να τα καταλάβω αυτά, ανέτρεξα στον Χόκμαν και στον Στρούμπελ Πέιτερ, ο οποίος είναι ένα είδος ε, Κάσπαρ, ήρωα, που λέει θα φάω τη σούπα. Αλλά η απάντηση είναι ότι όχι δεν θα φας τη σούπα, γιατί η Κομισιόν έχει βάλει στη σούπα τα λάθος συστατικά. Και καταλαβαίνετε και ξέρετε τι έγινε μετά από πέντε μέρες. Ο Κάσπαρ την έφαγε τη σούπα και πέθανε μετά από πέντε μέρες. Με λίγα λόγια, θέλω να πω ότι έχουμε ελαχιστοποιήσει τις ε, επιπτώσεις των συνεδριάσεών μας αυτής της Επιτροπής. Εδώ η ουσία είναι αυτό που υποσχέθηκε ο κύριος Γιούνκερ. Μια υπόσχεση όμως που δεν την τήρησε. Και εγώ θέλω να καταστήσω σαφές ότι οι διαδικαστικοί κανόνες ε, για τους τροποποιητικά μεταλλαγμένους οργανισμούς πρέπει να αναθεωρηθούν. Δεν θέλω η Επιτροπή να λάβει μια απόφαση κατά πλειοψηφία και αυτή είναι η ουσία του θέματος. Δηλαδή πρέπει να ζητήσουμε από τον κύριο Γιούγκερ να τηρήσει την υπόσχεσή του και όχι να κάνει αυτό που έκανε ο Κάσπαρ το γερμανικό παραμύθι που λέει όχι όχι εγώ δεν τη θέλω τη σούπα. Joy Flores, έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κοιτάξτε, εγώ διάβασα την αιτιολογία των αντιρρήσεων και ξεπλάγινε γιατί από ό,τι φαίνεται ότι υπάρχουν πολλοί που διαφωνούν με την αρχή που διέπει τους γενετικά τροπεπμένους οργανισμούς και συμφωνώ με την κυρία Παύλ ε, ότι ε, διαφωνεί γιατί είναι γενικά αντίθετη κατά των οργανισμών αυτών. Νομίζω ότι και η πράσινη είναι σαφής επ' αυτού και δεν το καταλαβαίνω αλλά δέχομαι τη θέση τους. Εκείνο όμως που δεν δέχομαι είναι το να υπάρχει ένα μείγμα αντισυντεχνιακό, λαϊκιστικό, που προβάλλουν διάφορα μέλη. Και εμείς ως σοσιαλδημοκράτες, οι Βρετανοί τουλάχιστον εργατικοί, εκπλήσονται που αναφέρεται εδώ ότι οι σοσιαλδημοκράτες ε, ε, στηρίζουν όλοι το θέμα αυτό. Εδώ ε, δεν ισχύει. Κάθε χώρα παίζει το δικό της εθνικό παιχνίδι και αυτό είναι ντροπή. Για μένα λοιπόν εδώ έχουμε να κάνουμε με μία ύπουλα απλουστευτική αντίρρηση και γίνεται αυτό διότι αυτός ο οργανισμός αντίσταται στο γλυφοσάτ που είναι ένα προϊόν που χρησιμοποιείται βρέως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα ε, χρησιμοποιείται σε 40% των ε, συγκομιδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που δεχόμαστε ε, είναι κάποιες εισαγωγές που χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν ε, και χρησιμοποιείται και το κάποιοι άλλοι βέβαια έχουν πρόβλημα με το γλυφοσάτ αυτό ε, γιατί είναι καρκινογενές ε, βεβαίως αυτό ισχύει Ισχύει το ίδιο και για άλλα προϊόντα, ίσως κάποια που ενέχουν, που έχουν μπέικον Έχουν λοιπόν, όπως σας είπα, μπέικον και θα πρέπει ίσως να συζητήσουμε και γι' αυτά. Είμαι όμως ε, προβληματισμένη, ακούω όλα αυτά που λέγονται εδώ. Έχουμε ένα σύστημα, το σύστημα αυτό λειτουργεί, ε, δόθηκε η δυνατότητα στους ευρωβουλευτές να απαγορεύσουν τις ζωοτροφές ε, από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και δεν το έκαναν. Το θέμα επανέρχεται από την πίσω πόρτα και είναι σαν να είμαστε στο σχολείο. Εντάξει, μπορεί κανείς να έχει τις αρχές του, αλλά θα πρέπει να ακολουθήσει τις σωστές διαδικασίες. Εδώ απλά ε, χάνουμε το χρόνο μας και γι' αυτό το λόγο εγώ δεν στηρίζω. Ευχαριστούμε. Ο Πρόεδρος. Δύο είναι ακόμα στον κατάλογο ο Μιλιτών και μετά κλείνει ο κατάλογος. πρώτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, νομίζω από αυτό το να στο NK6 ε, στο 603, ε, ίσως αυτό να μην είναι επικίνδυνο. Αλλά υπάρχουν άλλοι οργανισμοί που είναι ανθεκτικοί απέναντι στο γλυφοσάτ και ξέρετε τελικά αν καλλιεργείται ένα τέτοιο είδος αραβοσίτου στα δικά μας τα χωράφια, ενδέχεται οι γεωργοί να χρησιμοποιούν περισσότερο γλυκοσάτ. Άρα δηλαδή να χρησιμοποιείται περισσότερο αυτό το φυτοφάρμακο το γλυκοσάτ ε, στις δικές μας καλλιέργειες. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό το φυτοφάρμακο είναι επιβλαβές για την υγεία. Και δεν κατανοώ το γεγονός ότι εδώ στο Κοινοβούλιο δεν θέλουμε να αποκλείσουμε κινδύνους, έστω προληπτικά. Εγώ πιστεύω ότι προϊόντα που αυξάνουν τον κίνδυνο πρέπει να αποκλείονται. Και εδώ συμφωνώ με την προλαλή σας. Υπάρχουν σαφείς ε, κανονισμοί όσον αφορά τους ε, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και τα φυτά αυτά πρέπει να απαγορεύονται και εγώ λοιπόν συμφωνώ ότι καταβάλλονται προσπάθειες να εισαχθούν κάποια είδη από την πίσω πόρτα. Αυτό όμως δεν είναι σωστό. Δεν πρέπει να γίνεται πολιτική τέτοια μορφή. Ο τελευταίος στον καταλογό μου ε, είναι ο κύριος Μπάλτσα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να αντιδράσω ε, σε κάτι που ελέγχει σχετικά με τον κύριο Γιούγκερ ε, και τις υποσχέσεις που έδωσε. Και η πλειοψηφία των κρατών μελών όταν απορρίπτει τους ε, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, η Κομισιόν δεν θα πρέπει να δίνει την άδεια. Και όχι μόνο τον έφερε αυτό, στις προγραμματικές του δηλώσεις. Αυτό αναφέρεται και στο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν πρέπει λοιπόν να αυταπατάμετα. Ο πρόεδρος κ. Γιούγκερ είχε υποσχεθεί ότι δεν θα επιτραπεί κάτι τέτοιο και ανέφερε ότι η τροποποίηση του κανονισμού ε, η τροποποίηση αυτή θα εφαρμόζεται ε, και σε άλλους τομείς. Παναλαμβάνω λοιπόν, δεν πρόκειται μόνο για το ότι ο κύριος Γιούγκερ έδωσε μια υπόσχεση, αλλά και ο αρμόδιος επίτροπος είχε πει ότι η υπόσχεση αυτή δεν τηρείται. Και να πω και κάτι άλλο. Γιατί λέει η Επιτροπή ότι θα χορηγεί την άδεια αν δεν υπάρχει ειδική πλειοψηφία ούτε υπέρ ούτε κατά αυτού. Στην περίπτωση αυτή ούτε και η άποψη της ΕΦΣΑ είναι απορριπτική, άρα η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να δώσει την άδεια. Ε, θα πρέπει να μιλήσουμε για τη διαφάνεια όλων αυτών των ε, ενωσιακών οργανισμών. Ε, δεν ξέρω κατά πόσον υπάρχει ανεξάρτητος οργανισμός ο οποίος θα μπορούσε να τοποθετηθεί παράλληλα με την ΕΦΣΑ. Όσον αφορά στην ΕΦΣΑ γνωρίζουμε ότι πρόσφατα υπήρξαν παρεμφερή θέματα σε σχέση με βιοτεχνολογικά Ινστιτούτα και τον πρόεδρο της ΕΦΣΑ. Δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να δεχτούμε την παντοδυναμία της ΕΦΣΑ ή όχι. Πρόεδρος, Ευχαριστούμε. Τώρα, περιμένουμε σχόλια και απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ που δίνετε το λόγο στην Επιτροπή σχετικά με τα δύο αυτά ψηφίσματα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να υπενθυμίσω σε ποιο πλαίσιο ακριβώς βρισκόμαστε και γιατί συζητάμε τις προτάσεις αυτές. Εδώ αμφισβητείται το γεγονός, ε, το κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άσκησε τα εκτελεστικά της καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί και κατά πόσο τα έχει υπερβεί. Εδώ λοιπόν τη συζήτηση πρέπει να την βάλουμε στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Υπάρχει ρυθμιστικό πλαίσιο, υπάρχει διαδικασία το οποίο καταρτίστηκε από κοινού με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Και είναι αυστηρό. Όταν υπάρχει ένα αίτημα διοδότησης, εξετάζεται από την ΕΦΣΑ, την Ευρωπαϊκή μας Υπηρεσία δηλαδή ασφαλεία Τροφίμων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε δύο γεγονότα τα οποία διασταυρώθηκαν όσον αφορά το γενετικά τροπομένο αραβόσιτο δόθηκε έγκριση και μάλιστα ανανεώθηκε. Δεν πρόκειται για κάτι καινούριο. Παρ' όλα αυτά η ΕΦΣΑ κοίταξε κατά πόσο εφαρμόζεται το ΣΤΑΚ και διαπίστωσε ότι ο αραβόσιτος αυτός, ο γενικά το είναι εξίσου ασφαλής και κίνδυνος όσο και ο συμβατικός αραβόσιτος. Οι χώρες μέλη βέβαια υποβάλλουν σχόλια. Και άκουσα ότι κάποια σχόλια από τη Γαλλία, την Αυστρία και τη Γερμανία δεν λήφθησαν πλήρως υπόψη. Εδώ πρέπει να σας πω ότι εξετάστηκαν τα σχόλια αυτά από την ΕΦΣΑ και έφτασε σε διαφορετικό συμπέρασμα από ό,τι οι χώρες μέλη. Ή για κάποια άλλα χρειάστηκαν επιπλέον πληροφορίες και τελικά συμφώνησαν οι χώρες μέλη με το τελικό συμπέρασμα της ΕΦΣΑ. Η διαδικασία τώρα είναι ότι η γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ ε, παρουσιάσεται στο κοινό το οποίο είχε τη δυνατότητα να σχολιάσει. Κάτι το οποίο έγινε. Τα σχόλια πήγαν στην ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Τροφίμων και δεν βρήκε τίποτα από αυτά. Το επόμενο στάδιο της διαδικασίας, και σας το λέω για να καταλάβετε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο, στη συνέχεια όλα αυτά πήγαν ε, στην Επιτροπή των Χωρών Μελών και δεν υπήρξε καμία γνωμοδότηση από αυτή την Επιτροπή, δηλαδή δεν υπήρξε καμία πλειοψηφία ενισχυμένη ούτε υπέρ ούτε κατά. Επόμενο στάδιο της διαδικασίας είναι να πάμε στην Επιτροπή Έφεσης. Το ίδιο αποτέλεσμα. Δεν υπήρξε γνωμοδότηση ούτε υπέρ ούτε κατά. Τι συμβαίνει λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις. Η απόφαση για την επιτροπολογία είναι σαφή. Εφόσον δεν υπάρχει γνωμοδότηση, ούτε κατά, ούτε υπέρ, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το μέτρο. Μπορεί να εγκρίνει το μέτρο. Εδώ για τους γενικά δομημένους οργανισμούς υπάρχει το δικαίωμα για τον αναφέροντα να έχει απάντηση στο αίτημά του για διοδότηση. Εμείς πιστεύουμε ότι εδώ δεν υπερβήκαμε τα εκτελεστικά μας καθήκοντα και ότι τηρήσαμε απόλυτα τις διαδικασίες. Τώρα, βέβαια, Καταλαβαίνετε τη συζήτηση που κάνετε εδώ, όπου εκφράζεται απογοήτευση για την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υποσχέθηκε ο πρόεδρος Γιούγκερ Δεν προχωράει περισσότερο. Ακούσατε τον Επίτροπο στην Ολομέλεια που εξήγησε για ποιο λόγο πιστεύουμε ότι όπως οι χώρες μέλη στην ψηφοφορία, κάποιες τουλάχιστον, λένε ότι δεν θέλουν να δώσουν την άδεια σε κάποιο προϊόν ή θέλουν να απόσχουν για άλλους λόγους, όχι για λόγους επιστημονικούς. Γι' αυτό και η Επιτροπή τελικά πρότεινε το κείμενο αυτό για την καλλιέργεια, με το οποίο επέτρεψε στις χώρες μέλη να αρνηθούν την άδεια για λόγους άλλους πλην επιστημονικούς είτε πρόκειται για κοινωνικού λόγους, είτε για οτιδήποτε. Θελήσαμε να δώσουμε το δικαίωμα αυτό στις χώρε μέλη και αυτό ακριβώ προτείναμε στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Το δικαίωμα αυτό τώρα δεν επιβλήθη στο Κοινοβούλιο. Θα βοηθούσε τις χώρε μέλη που λένε ότι δεν θέλουμε αυτό τον, μη, τον γενετικά δομένο οργανισμό όχι για λόγους επιστημονικούς αλλά για άλλους. Ο Επίτροπος είπε ότι δεν θα επανέλθουμε με άλλη πρόταση. Δεν υπάρχει σχέδιο Β. Έχουμε μόνο το σχέδιο Α, που είναι η πρόταση που έχετε. Και δεν έχει πεθάνει ακόμα αυτή η πρόταση, παραμένει, εφόσον ε, συζητιέται και σε επίπεδο Συμβουλίου σύντομα. Και όπως είπε ο Επίτροπος, είναι μια συζήτηση σίγουρα χρήσιμη και σημαντική, γιατί μας κάνει να αντιληφθούμε ότι υπάρχει μια διαφορά είτε είναι ο Γενικό Διευθυντής είτε ο κύριο Λάστικο που ήρθε εδώ, το λένε και το ξαναλένε, οι χώρες μέλη έχουν μία θέση στην ψηφοφορία και μία διαφορετική όταν πρόκειται για τη χρήση. Η πρόταση αυτή λοιπόν παρατείνει τη συζήτηση, κάτι το οποίο είναι προς όφελος όλων και τη Επιτροπής και του Κοινοβουλίου και των πολιτών, γιατί έτσι καταλαβαίνουν ακριβώς τι γίνεται και ποια είναι η θέση των κρατών μελών και των υπολείπων. Συνοψίζοντας, πιστεύουμε ότι δεν έχουμε υπερβεί τα εκτελεστικά μας καθήκοντα ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτείνοντας για ψηφοφορία το γενετικά αυτό τροποποιημένο αραβόσιτο. Πρόεδρος. Ωραία. Αν όσοι έχουν υποβάλει τι αντιρρήσει ενστάσει θέλουν να παρέμβουν, παρακαλώ και σύντομα, γιατί μα πιέζει κάπω ο χρόνο. Ο κύριο Σωστά. Θα είμαι σύντομο. Γιατί και εγώ πρέπει να πάω στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού, γιατί έχω μια άλλη έκθεση εκεί. Για τον κύριο Φιένερ. Κοιτάξτε. Να κάνουμε όπως κάποιοι αρνούνται την κλιματική αλλαγή και να αρνούμεθα επιστημονικές απόψεις, ε, νομίζω ότι είναι τραβηγμένο από τα μαλλιά. Έχουμε τη γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ, το εξηγήσαμε, και της Διεθνούς Υπηρεσίας για την έρευνα στον καρκίνο και πρέπει να συγκρίνουμε αυτές τις δύο αυτά τα δύο κείμενα, αυτές τις δύο μελέτες έχουν βέβαια διαφορετική μεθοδολογία και διαφορετικά πράγματα ψάχνουν. Σήμερα το μεσημέρι έχω μία συζήτηση όπου και ο, Επίτροπο, και ο Πρόεδρος της ΕΦΣΑ και ο κύριος Γιάκ θα έρθουν στο κτίριο της ε, Δυτικής Φλάνδρας και θα έρθουν εκεί να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα. Ο φιλελεύθερος συνάδελφος από τη Σουηδία υπογράμμισε ότι η πραγματική συζήτηση είναι, και το είπαν και άλλοι, ότι ο κύριος Γιούγκερ δεν τηρεί τις υποσχέσεις του. Πάνω σε αυτό πρέπει να επιμείνουμε. Και με το κείμενο αυτό μπορούμε να πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι θετικό αυτό για να τηρούν τις υποσχέσεις τους. Να έρθουν με μια σοβαρή πρόταση. Γιατί έτσι θα το λάβει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλες τις, τις προτάσεις. Νομίζω λοιπόν ότι όντως πρέπει να επιμένουμε και να πιέσουμε την Επιτροπή γι' αυτό. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Τέλος. Η κυρία τον Άνω που εκπροσωπεί την κυρία Κοντονίν. Εκτός μικροφώνου δεν την ακούμε, την κυρία Τον Τονάνο. Α, ναι, ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα σε αυτά που υπόθηκαν. Πρόεδρος, θα ψηφίσουμε στις 4 το απόγευμα. Τον Ιανουάριο θα πάει στην Ολομέλεια. Περνάμε στο σημείο 9. Ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τον έλεγχο καταλληλότητά στον τομέα δίλησης πετρελαίου. Θα δώσω το λόγο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Κάρλο Πετινάρη. Η Γενική Διευθύνση Growth. 10 λεπτά με ένα τέταρτο, καλύτερα 10 λεπτά παρά 15. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Good morning. Um, Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Εγώ δεν είμαι ο Πετινέλη, είμαι ο Μπίσο. Ο κύριος Πετινέλη είχε να πάει κάπου αλλού. Α, όχι, νάτος, νάτος. Όχι, λάθος, ε, έρχεται, οπότε επιτρέψτε μου να του δώσω και το λόγο. has the floor, please.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 λυπάμαι που καθυστέρησα, αλλά τελικά καθυστέρησα περισσότερο στον έλεγχο ασφαλείας από ό,τι είχα υπολογίσει. Αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πάρα πολύ ε, που με προσκαλέσατε σήμερα εδώ και μου δίνετε τη δυνατότητα να σας εξηγήσω πώς έχει η κατάσταση όσον αφορά το fitness check, τον έλεγχο πεπραγμένων σχετικά με τα δηληστήρια και την δήληση πετρελαίου. Ε, πρώτα απ' όλα ε, να σας πω ότι υπάρχει μία μελέτη που έγινε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία ε, αναφέρει τον, ε, το θέμα του ελέγχου καταλληλότητας. Μόλις γίνει ο έλεγχος καταλληλότητας βρισκόμαστε πια στην τελευταία φάση προετοιμασιών δεν μπορώ να δεσμευτώ για συγκεκριμένη μέρα, αλλά πια μιλάμε για κάποιες εβδομάδες μέχρι να ολοκληρωθεί το θέμα. Και όσον αφορά λοιπόν τον έλεγχο καταλληλότητας και τη σχετική μελέτη, η μελέτη αυτή θα δημοσιευτεί στο διαδίκτυο και βέβαια είναι σαφές, θα αποσταλεί ε, στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Όλα αυτά γίνονται για να αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις της ε, νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα δίλης πετρελαίου. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ ελέγχου καταλληλότητας και μια κλασικής μελέτης επιπτώσεων, η οποία η τελευταία εστιάζεται στις επιπτώσεις μιας συγκεκριμένης πρότασης, αλλά η δικιά μας αφορά τις επιπτώσεις όλης της νομοθεσίας, του συνόλου των νομοθετικών πράξεων. Επιλέξαμε λοιπόν τον ε, τομέα διήλυσης πετρελαίου για τον έλεγχο καταλληλότητα, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε, αυτό είναι κάτι από τα πρώτα που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια δεν θα είναι και το τελευταίο που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προχωρήσει περαιτέρω στο θέμα των ελέγχων καταλληλότητας. Αυτό που μας ενδιέφερε, ο λόγος που έγινε ως πρώτος έλεγχος, ήταν ότι υπάρχει μια ομοιογένεια ο δεύτερος λόγος είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη το 2012 είχε αναφέρει ότι δεν θα ήταν σκόπιμο να ελέγξει κανείς ε, την τρέχουσα νομοθεσία για επιπτώσεις ε, ε, στην ανταγωνιστικότητα κυρίως του ελέγχου του τομέα δίλης πετρελαίου, γιατί υπάρχουν όλο και περισσότερο δηληστήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χάνονται θέσεις εργασίας. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να υπάρχει ασφάλεια εφοδιασμού. Από το 7 13 σε 13 δηληστήρια της Ευρωπαϊκής που έκλεισαν, εκεί έγινε έλεγχος καταλληλότητας και αυτό οδήγησε στο ότι χάθηκαν άμεσα 10.000 θέσεις εργασίας και τουλάχιστον 40.000 θέσεις εργασίας έμεσα. Έτσι λοιπόν το έγγραφο ε, θα είναι ο έλεγχος καταλληλότητας που έχουμε κάνει και αυτό θα παρουσιάζει μια ε, ολιστική προσέγγιση του πώς διάφορες νομοθετικές πράξεις επηρεάζουν ένα συγκεκριμένο οικονομικό τομέα. Ε, η στρατηγική καλύτερη νομοθεσία οδηγεί σε ελέγχου καταλληλότητα και σε αναθεώρηση τη νομοθεσία, κυρίω των επιπτώσεών τη. Και αξιολογείται η αποτελεσματικότητα, η συνοχή, αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στην ανάλυση τη ανταγωνιστικότητα του τομέα. Η ανάλυση της, που γίνεται στην έκθεση είναι αναδρομική και εστιάζεται στον τομέα δίλης πετρελαίου κατά την περίοδο 2000 2012. Αυτό λοιπόν το έγγραφο εργασίας είναι ένα έγγραφο το οποίο προέκυψε από το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η επιλογή των μέτρων έγινε ανάλογα με τη σημασία των τομέων μετά από διαβουλεύσεις και πριν εγκριθεί η εντολή για τον έλεγχο καταλληλότητας. Η ποσοτική αξιολόγηση έλαβε υπόψη της τις επιπτώσεις της νομοθεσίας, το κόστος και ε, στην ε, βιομηχανία πετρελαίου γενικότερα. Στόχος είναι να παραμείνουμε διεθνώς ανταγωνιστικοί. Η νέα νομοθεσία εντοπίζει για τον τομέα κάποια μέτρα όπως οδηγία για τις ενώσεις πηγές ενέργειας, ε, η οδηγία περί ανταλλαγής ποσοστώσεων εκπομπών, η οδηγία περί βιομηχανικών εκπομπών ε, και άλλα μέτρα. Όσον αφορά το κόστος και το όφελος, το μέσο κόστος ε, στην περίοδο 2000-2012 ε, είναι αναλογικό σε σχέση με τα ωφέλη. Παρόλα αυτά, το μέσο σωρευτικό κόστος των νομοθετικών πράξεων δεν είναι αμεληταίο και υπολογίζεται στο 25% σε σχέση με τη μείωση του καθαρού περιτορίου κέρδους. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες ε, και επηρεάζουν την οικονομική απόδοση του τομέα διήλυσης πετρελαίου. Όσον αφορά αυτούς τους άλλους παράγοντες, μερικοί είναι πολύ εξειδικευμένοι στα δηληστήρια, ας πούμε μέγεθος του δηληστηρίου ε, και παρεμφερία. Άλλοι παράγοντες όμως περιλαμβάνουν το σχετικά υψηλό επίπεδο διαφοροποίησης, κυρίως το ενεργειακό κόστος ε, και τη διαθεσιμότητα των ε, προϊόντων πετρελαίου που παράγουν τα δηληστήρια. Αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση δουλεύουν για μια παγκόσμια αγορά. Όσον αφορά τον ανταγωνισμό ανάμεσα στα ευρωπαϊκά δηληστήρια και αυτά από κάποιες άλλες περιοχές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Νοτιοανατολική Ασία, η αυστηρή εφαρμογή των περιβαλλοντικών κανόνων, αυτή ισχύει για όλους. Παρόλα αυτά, αυτό δεν ισχύει για ανταγωνιστές από την πρώη Σοβιετική Ένωση και τη Μέση Ανατολή. Επιπλέον, τα μεγάλα δηληστήρια στη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία έχουν χαμηλότερο ενεργειακό κόστος. Ε, η ίση όρια ανταγωνισμού με τρίτες χώρε είναι καθοριστικό για να λειτουργεί κανεί σε μια παγκόσμια αγορά. Τα δηληστήρια όχι μόνο παράγουν προϊόντα, αλλά είναι σημαντικά και για άλλες μεταποιητικές ε, βιομηχανίες. Το πρώτο λοιπόν αποτέλεσμα της ανάλυσης μας δεν δείχνει να υπάρχει επικάλυψη ή ασυνέπειες στη νομοθεσία του αντίον ε, διαπιστώνονται συνέργειες, κυρίως έχοντας κατά νου τις υποχρώσεις αναφοράς με βάση τη σχετική νομοθεσία. Ε, στην περίοδο, κατά την περίοδο που μελετήσαμε, διαπιστώσαμε ότι το ρυθμιστικό κόστος αυξήθηκε από το 2000 μέχρι το 2008 και μετά το 8 μοιάζει να έχει μέχρι το 2012. Εντοπίσαμε τις επιπτώσεις του κανονισμού στο κόστος της απόδοσης των δηληστήρων, αλλά αυτό βέβαια εξαρτάται σε κάποιο βαθμό και από τις επενδύσεις και τα πάγια έξοδα γιατί σε άλλες περιπτώσεις έχουν γίνει προσαρμογές καλύτερο ανταγωνισμό. Τα πιο αποτελεσματικά δηληστήρια μπόρεσαν να απορροφήσουν το κόστος και να παραμείνουν επικερδοί, αλλά δεν ισχύει αυτό για όλα τα δικαστήρια. Ε, γενικά λοιπόν, και τώρα θα σας αναφέρω ε, κάποιο σημαντικό στοιχείο, 47 σεν το βαρέλι είναι το, η μέση παραγωγή, η οδηγία ε, για τις εκπομπές κοστίζει 13 cent και η άλλη ε, για τις ανώσιμες πηγές 3,7 cent. Θα ήθελα τώρα να εστιάσω την προσοχή μου σε κάποιες παρατηρήσεις που αφορούν σε μεμονωμένες νομοθετικές πράξεις. Οι μεμονωμένες νομοθετικές πράξεις μπορούν να επηρεασούν τις επιπτώσεις μιας οδηγίας, μπορούν να αλλάξουν οι προδιαγραφές. Και ένα από τα σημαντικότερα ωφέλη που προκύπτουν από την οδηγία ε, περί ενώσεων πηγών ε, και ε, φορολογίε είναι η ανεξαρτητοποίηση δίζελ από τη Ρωσία. Αυτό οδήγησε στο να υπάρχει ανεξαρτητοποίηση από 1 μέχρι 6,3% αλλά παρόλα αυτά ε, θέλω να επισημάνω ότι πρόκειψαν και κάποια άλλα έσοδα ε, για τα δηληστήρια 3,7 σέντα αναβαρέλι ε, αργού πετρελαίου. Στις πρώτες δύο εμπορικές περιόδους διαπιστώνουμε ότι υπήρχε επιβάρυνση τομέα και αυτό δεν σημαίνει απλά ότι όλα τα δηληστήρια επιβαρύνθηκαν ιδιαίτερα, ε, η κατάσταση ποικίλει. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να πω ότι δεν πρόκειται για ένα ιδιαίτερο μειονέκτημα της οδηγίας περί ποσοστώσεων. Εμείς πιστεύουμε ότι η επιβάρυνση ε, μπορεί να εξηγηθεί με την μεγαλύτερη επιβάρυνση και με χαμηλότερο επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας. Οι δύο λοιπόν οδηγίες που οδήγησαν σε μεγαλύτερη αύξηση του κόστους παραγωγής ήταν η οδηγία περί βιομηχανικών εκπομπών ε, και η οδηγία περί ποιότητας καυσίμων. Η πρώτη κόστισε 5 εκατομμύρια ευρώ κεφαλαιοχικών επενδύσεων αναδηληστήριο. Αυτό αυξήθηκε το ποσό μετά το 2006 και συνδέθηκε πάγιες δαπάνες 1,8 δις ευρώ σε τήσια βάση αναδηληστήριο. Οι οικονομικές επιπτώσεις της οδηγίας περιποιότητας καυσίμων σε μεγάλο βαθμό συνδέεται και με άλλες διατάξεις που όμως δεν οδήγησαν σε ε, χειροπιαστά αποτελέσματα. Ας δούμε λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε το αποτέλεσμα του ελέγχου καταναλώτε θα είναι κρίσιμο για να χαράξουμε πολιτική. Το επόμενο σχετικό φόρουμ προβλέπεται για την 1η Μαρτίου του 2016 στις Βρυξέλλες. Εκεί θα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι άμεσα εμπλεκόμενοι, θα αποτελεί ορόσημο όπου θα συζητηθούν τα αποτελέσματα του ελέγχου καταλληλότητας για τα δηληστήρια. Αυτό ο έλεγχος καταλληλότητας θα είναι ένα εργαλείο μεταξύ άλλων νομοθετικής και μη νομοθετικής φύσεως, όπως είναι αξιολόγηση ε, κόστος, αξιολόγηση σωρευτικού κόστου και ούτω καθεξής. Ε, τα αποτελέσματα του ελέγχου καταλληλότητας είναι πολύ ευρύτερα από, ε, από την μελέτη αντικτύπου, γιατί όπως σας είπα η δεύτερη αφορά μεμονωμένες νομοθετικές πράξεις ο έλεγχος καταλληλότητας και τα αποτελέσματά του θα στηρίξουν και την αναθεώρηση της επερχόμενης ε, νομοθεσίας. Εδώ για τα δηληστήρια έχουμε πολύ καλή νομοθεσία, λαμβάνει υπόψη στο περιβάλλον. Θεωρούμε λοιπόν ότι δεν πρέπει να χάσουμε αυτό το στοιχείο είναι απαραίτητο να υπάρχει μια ισχυρή νομοθετική βάση για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σημαντικούς περιβαλλοντικούς στόχους και να αυξήσουμε παράλληλα και τις θέσεις απασχόλησης. Είναι λοιπόν όλο καθοριστική σημασία για να επιδιώξουμε επιτυχία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Το λόγο η κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ Μπορούμε να ευχαριστήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση που ακούσαμε και την τεράστια εργασία που έκανε διότι ο έλεγχος καταλληλότητας είναι ένας πολύ σωστός τρόπος για να προχωρήσουμε στην αξιολόγηση και την επίπτωση της νομοθεσίας σε έναν ε, βιομηχανικό κλάδο. Αλλά όταν κάνουμε αυτού του είδους τον ε, απολογισμό δεν θα πρέπει να παραμείνει είναι πρόγραμμα, θα πρέπει να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα. Λοιπόν, αυτός ο έλεγχος καταλληλότητας στον τομέα της διήλυσης δείχνει την έκθεση του τομέα στην στον εξωτερικό ανταγωνισμό, αυτό που καταστεί, την Ευρώπη ιδιαίτερα ευαίσθητη και ευάλωτη. Αυτό που έχει σημασία είναι να γνωρίζουμε ο πλευράς Κομισιόν εάν προτίθεται να λάβει μέτρα και πια για την διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου, να περιοριστούν τα επιπλέον, επιπλέον δαπάνες και μας είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει επανεξέταση κάποιων νομοθεσιών, τι προβλέπει λοιπόν, πώς και ούτω καθεξής. Έπειτα η Κομισιόν μπορεί να μας πει τα μέτρα τα οποία προβλέπονται στο πλαίσιο του OTS για το ζήτημα της δίλησης πετρελαίου, διότι ξέρουμε ότι έχουμε χάσει πολλά δηληστήρια και άρα πολλές θέσεις απασχόλησης και τα δηληστήρια που έχουμε στην Ευρώπη Ακόμα και αν διατηρούμε την πρώτη θέση σε επίπεδο ποιότητα, δυστυχώ βαίνουν μειούμενα. Και τελευταία ερώτηση θα θέλω να γνωρίζω αν η Κομισιόν προβλέπει να μα μιλήσει για την συνέχεια αυτού του ελέγχου καταλληλότητα ε, σε τακτά διαστήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. για να συγχαρώ πρώτα απ' όλα την συνάδελφο που μίλησε πριν από μένα αλλά και την Κομισιόν και να ζητήσω ότι αυτός ο έλεγχος καταλληλότητας ε, να μην εγκαταλειφθεί αλλά να συνεχιστεί να, αποτελεί, να συνεχίσει να αποτελεί μια βάση για την ε, επιπτώσει ε, των νέων ρυθμίσεων των μέτρων αγωνιστικότητας του κλάδου που ακόμα και σήμερα σε όλες τις μελέτες σχετικά με το ενεργειακό μείγμα έχει ιδιαίτερη σημασία τουλάχιστον μέσω πρόθεσμα. πέραν του ότι ο χρόνος που έχει ληφθεί υπόψη ε, φτάνει μέχρι το 2012 αλλά υπάρχει και το μέλλον έχω υπόψη μου το OTS και το κόστος που προκαλείται για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ενώ οι επιχειρήσεις εκτός Ευρώπης δεν έχουν τέτοιο, παρόμοιο κόστος, παρόμοιες δαπάνες. Θα υπάρχουν λοιπόν επιχειρήσεις οι οποίες θα ευαρεθούν περαιτέρω. Θα ήθελα να γνωρίζω λοιπόν από την Κομισιόν πώς και πότε θα τα συμπεριλάβει στην αξιολόγησή της. Επίσης θα ήθελα να μάθω όταν αναφέρεται ότι υπάρχουν δηληστήρια που έχουν ε, εντάξει το, τις δαπάνες αυτές παραμένοντας ανταγωνιστικές, θα ήθελα να μάθω πόσες, είναι αυτά τα δηληστήρια επί του συνόλου που μπόρεσαν να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητα και μπόρεσαν να απορροφήσουν αυτές τις δαπάνες. Πώς το πέτυχαν, διότι τα δηληστήρια μπορούν να ε, μετακυλήσουν το κόστος τους ε, καταναλωτές. Είδαμε ήδη μελέτες που μας το αναφέρουν, αλλά και εδώ οι επιπτώσεις είναι χάσιμο ποσοστών στην αγορά και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί και να μας εξηγηθεί καλύτερα από την Κομισιόν. Επίσης ε, κρίνω πως χρειάζεται να εξετάσουμε αυτή τη συνολική κατάσταση. Είναι κάτι το οποίο θα αντιμετωπίσουμε στο εγγύς μέλλον και μπορεί να οδηγήσει από επενδύσεις στην Ευρώπη διότι το υψηλότερο κόστος το έχει αναγνωρίσει η Κομισιόν δεν είναι 0,41 cents ανά Βαρέλη, αλλά εάν εμεί μεταφέρουμε τις, ε, την παραγωγική ικανότητα σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, από όπου η Ευρώπη θα συνεχίσει να εισαγάγει, διότι το ζήτημα ενδιαφέρει την οικονομία μας, εμείς θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα το, οποίο οδηγεί στην απώλεια θέσεων απασχόλησης, αύξηση του ενεργειακού κόστου και ούτω καθεξή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω να ρωτήσω κάτι την Επιτροπή όσον αφορά το όλο αυτό το θέμα. Αναρωτιέμαι κατά πόσο μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζονται για θέματα που έχουν να κάνουν ε, με την ε, δίληση ανατομέα. Εμείς εξετάζουμε ε, το θέμα της απασχόλησης. Σίγουρα παίζει ρόλο εδώ. Πρέπει να δούμε και το θέμα του περιβάλλοντος, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τεράστιες προκλήσεις δηλαδή που έχουμε μπροστά μας. Όμως το ερώτημα είναι, οι χώρες μέλη τι κάνουν για να χρησιμοποιήσουν περισσότερο νέες τεχνολογίες και νέα καύσιμα. Και αυτά τα νέα καύσιμα πώς στηρίζονται ώστε να έχουμε στο μέλλον καύσιμα τα οποία να προστατεύουν το περιβάλλον και να μην το καταστρέφουν. Αναρωτιέμαι λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση τι δουλειά κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. δημιουργεί ανταγωνισμό για καλύτερη χρήση καυσίμων στις μεταφορές ώστε η δήληση πετρελαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει και ανταγωνιστική αλλά και φιλική προς το περιβάλλον. Ωραία, πολλές οι ερωτήσεις, ίσως η Επιτροπή να έχει να απαντήσει κάτι σε όλα αυτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Για την κυρία Ρουσπέ και όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και τι σκοπεύουμε να κάνουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως είπα και πριν στην παρουσίασή μου, θα υποβάλει τον έλεγχο καταλληλότητας. Σήμερα δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα κάνουμε, όχι γιατί δεν έχουμε ιδέες, αλλά γιατί θέλουμε πρώτα να συγκρίνουμε τις ιδέες μας πρώτα απ' όλα με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αλλά και με την κοινωνία των πολιτών και με την βιομηχανία και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Πρώτα θα έχουμε τα φόρουμ με τον κλάδο της δίλησης πετρελαίου και όλους τους ενδιαφερόμενους του κλάδου. Από εκεί και πέρα, προς το παρόν δεν έχω πληροφορίες για τα αποτελέσματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κάνει το fish τσέκ check για κάποιους τομείς. Τώρα τον έλεγχο αυτό καταλληλότητας τον κάνουμε για τη δίληση πετρελαίου. Δεν ξέρω κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει και σε άλλους τομείς. Δεν προβλέπεται προς το παρόν, αλλά δεν αποκλείεται. Μπορεί. Για την κυρία Γκαρντίνη, η Κομισιόν φυσικά συμφωνεί απόλυτα πως ε, ο αντιγωνιστικό της τη βιομηχανία πετρελοειδών έχει ιδιαίτερη σημασία. Πρέπει να εγγυηθούμε το ενεργειακό μείγμα. διότι όπως είπα και στην παρέμβασή μου η βιομηχανία διήλυσης παράγει και άλλα προϊόντα για την, ε, με, τη βιομηχανία τη μεταπαιδική και ως εκ τούτου είναι σημαντικό για όλη την αλυσίδα παραγωγής. Είναι γεγονός ότι η μελέτη καλύπτει την περίοδο 2000-2012. Από το 2012 και μετά υπήρξαν διάφορες αλλαγές, αλλά όπως είπα, απαντώντας και στην προηγούμενη ε, συνάδελφό σας, η Κομισιόν δεν έχει προγραμματίσει ε, περαιτέρω ενημέρωση και επικαιροποίηση της μελέτης. Αυτό που έχει σημασία είναι να παρουσιαστεί η μελέτη αυτή στις αρχές του 2016, να κάνουμε ένα απολογισμό της αποτελεσματικότητας και της προσθέμενης αξίας της και μετά θα ε, δούμε ε, ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Τώρα σε ό,τι αφορά ποια δηληστήρια μπόρεσαν να απορροφήσουν τον δαπάνη αυτή. Αυτό ίσως περιλαμβανθεί στη μελέτη που θα δημοσιευθεί. Προς το παρόν δεν έχω αυτή τη δημοσίευση, αλλά προς το παρόν τους παράγοντες τους ανέλησα στην παρανομιλία μου. Αυτό εξαρτάται από την τεχνολογική πρόοδο, από την από το δηληστήριο, το κόστος διήλυσης για ένα δηληστήριο είναι ένα κόστος ιδιαίτερα υψηλό και σημαντικό. Όλοι αυτοί είναι παράγοντες οι οποίοι συνέβαλαν στο να διατηρηθούν κάποια δηληστήρια πιο ανταγωνιστικά ενώ άλλα δεν το επέτυχαν. Σε ό,τι αφορά την μεταφορά του κόστου, τη μεταχείριση του κόστου στους καταναλωτές. Αυτό είναι κάτι το οποίο έγινε αντικείμενο πολλών συζητήσεων, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της οδηγίας ETS ε από ό,τι γνωρίζω δεν υπάρχουν μελέτες ε, που να δίνουν τελικά συμπεράσματα. Υπάρχουν διάφορες ε, υποθέσεις, ε, μελέτες κλπ. Δεν υπάρχει απόδειξη ότι κάποια μελέτη είναι πιο σωστή από άλλες. Πάντως πρόκειται για κόστη στο οποίο μετακυλείται σε άλλους δεν είναι κόστος, το κόστος τα οποία απορροφώνται και δεν είναι κάτι το οποίο κάνει τις ε, βιομηχανίες αυτές να ε, χάσουν ανταγωνιστικότητα. Ε, συνήθως πρόκειται για ιδιώτες καταναλωτές, πρόκειται τους πολίτες με λοιπόν, το κοιλία δεν το κόστος. Άρα δεν είναι ένα στοιχείο, το οποίο μπορούμε να εξετάσουμε εύκολα. Επαναλαμβάνω μόνο ότι υπήρξαν πολλές μελέτες, δεν υπάρχουν συμπεράσματα ε, ε, ε, ένα κίνδυνο σε ό,τι αφορά την αποεπένδυση στην Ευρώπη, φυσικά η Κομισιόν γνωρίζει και προσπαθεί με κάθε τρόπο να αυξήσει τι επενδύσεις στην Ευρώπη. Παράδειγμα, το σχέδιο, επενδυτικό σχέδιο 315 δις ευρώ είναι ένα παράδειγμα σαφές αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι οι επενδύσεις για τις μεγάλες πολυεθνικές οι οποίε θα πρέπει να αποφασίσουν οι πολυεθνικέ το πού θα κάνουν τις καταθέσεις, τις επενδύσεις τους, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που υπάρχει ανάπτυξη, αν λοιπόν σε άλλες περιοχές του κόσμου υπάρχει ανάπτυξη πιο δυνατή, πιο ισχυρή, οι μεγάλες πολυεθνικές που δρούν παγκοσμίω έχουν την τάση να επενδύουν σε αυτές τι καταθεσεις του επενδυσεις διότι απο πολλου παραγοντε υπάρχει μεγαλύτερη ανάπτυξη και έτσι είναι δύσκολο οι μεγάλε είναι αντιμετωπίσουμε αυτή την τάση με τεχνικές ε, ε, λύσεις. Το σχετικά με την τρίτη παρέμβαση και θα ολοκληρώσω πώς πιστεύουμε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε με τον βιομηχανικό κλάδο. Φυσικά συνεργαζόμαστε με τον κλάδο αυτής εξ αρχής αυτής της δραστηριότητας ε, ελέγχου καταλληλότητας. Πριν να ξεκινήσει λοιπόν αυτή η προσπάθεια έγινε διαβούλευση τεχνική έκθεση που προετοιμάζει το Κοινό Κέντρο Ερευνών και πιο, ακόμη πιο σημαντικό θα είναι ότι θα υπάρξει μια ανοιχτή ζήτηση την 1η Μαρτίου εδώ Βρυξέλλες με όλους τους ενδιαφερόμενους, τα δηληστήρια, την βιομηχανία, ε, μη κυβερνητικού οργανισμούς και όλους όσοι θα θελήσουν να συμμετάσχουν, ελπίζω να υπάρξουν κάποια μέλη από το Ευρωκοινοβούλιο. Φυσικά Γνωρίζουμε ότι ο τομέας της διήλυσης κατά κάποιο τρόπο ανταγωνίζεται με άλλες πηγές ενέργειας ε, στο των μεταφορών. Η Κομισιόν έχει μια στρατηγική για τις αναλλακτικές καύσιμα για μεταφορές και τα προϊόντα της ε, διήλυσης είναι ένας από τους τρόπους αυτούς. Υπάρχει και ο αλλά για το ζήτημα αυτό υπάρχει μια ειδική στρατηγική που νομίζω βρίσκεται υπό την ευθύνη του αρμόδιου επιτρόπου για τις μεταφορές. Αυτά είχα να πω, αλλά ε, ο εμπειρονούμενος μου και εγώ θα παραμείνουμε στη διάθεσή σας, αν υπάρχουν ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή συζήτηση. Το επόμενο θέμα στην μέση διάταξη είναι πολύ σοβαρό και περιμένουμε ακόμα τους προσκεκλημένους μας. Γι' αυτό για ένα τέταρτο θα σταματήσουμε και θα περάσουμε μετά στο σημείο 10 που είναι η ανταλλαγή απόψεων με τον ΠΟΕ και την ΕΦΣΑ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την ουσία γλυφοσάτ. Honorable colleagues, I just want to inform you that uh, people from IR are already in the premises of European Parliament. But... Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι οι προσκεκλημένοι μας εδώ, αλλά κάτω στην ασφάλεια στους ελέγχους. Οπότε θα πάρει άλλα πέντε λεπτά. Πέντε λεπτά λοιπόν ακόμα διάλειμμα. Dear colleagues, it is... Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να αρχίσουμε πια. Με το θέμα 10 που είναι η ανταλλαγή απόψεων με τον ΠΟΕ, την ΕΦΣΑ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την ουσία glyphosate. Έχουμε, έχουμε εδώ λοιπόν τον ΠΟΕ, την ΕΦΣΑ, την Επιτροπή. Υπάρχει η μελέτη και θα δώσω το λόγο στον δόκτορα Κρίστοφερ Βάιλτ που είναι της CRC και τον κύριο Ούτροκ που είναι υπεύθυνο για το γλυφοσάιτς υποθέτω και μετά θα έχουμε τον πρόεδρο και τους εμπειρογνώμονες της ΕΦΣΑ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Ξέρω ότι έχουμε λίγο χρόνο Οπότε θα σας παρουσιάσω την Kate Guyton που θα αναφερθεί στην αξιολόγηση των δεδομένων. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Πολύ χαίρομαι που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας. Μέσα στα επόμενα 10 λεπτά, 15, θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω όχι μόνο πώς γίνεται η αξιολόγηση βάσει του μονογραφικού προγράμματος, αλλά και ποια ήταν τα αποτελέσματα για το γλυφοσάτ. Αλλά δεν ξέρω πώς να προχωρήσω τις διαφάνειες, λέει η Μιλήτρια. Great. So Ωραία. Θα σας δώσω το πλαίσιο όσον αφορά τα μονογραφικά προγράμματα και τις ταξινομήσεις και μετά θα μιλήσουμε για τις αξιολογήσεις του Glycosat. Η οργάνωσή μας ε, είναι 50 ετών και πριν υπήρχε η ιδέα να δημιουργήσουμε ένα σύστημα ταξινόμησης για τις καρκινογενείς ουσίες. Το πρόγραμμα αυτό γεννήθηκε λοιπόν υπό το Λορέντσο Τομάτης. Βλέπετε τη φωτογραφία του στη διαφάνεια. Η ιδέα του ήταν ότι θα μπορούσε να υπάρχει μια συστηματική αξιολόγηση και στοιχεία με επιστημονικά δεδομένα για τις καρκινογενείς ουσίες. Και βάσει αυτής της ιδέα συνεχίζουμε και εμείς. Τα τελευταία, τα τελευταία λοιπόν 40 χρόνια αξιολογήσαμε πάνω από 980 παράγοντες. Ο λόγος που γίνονται οι συστάσεις έχουν να κάνουν και με την έκθεση, αλλά και κυρίως με το πόσο καρκινογενείς είναι οι παράγοντες αυτής. Οπότε έχουμε κάποια το οποίο θεωρούμε ότι δεν είναι καρκινογενή, αλλά υπάρχουν και άλλες που δεν μπορούμε καν να ταξινομήσουμε στην κατηγορία 3. Κάποιοι παράγοντες ταξινομούνται στην ομάδα 1, μετά έχουμε την ομάδα 2α και την ομάδα 2β. Ότι τα στοιχεία μας χρησιμοποιούνται από διάφορους ε, αξιωματούχους σε χώρες μέλη που ασχολούνται με την υγεία για να προστατεύσουν καλύτερα τον πληθυσμό. Εδώ λοιπόν θα αναρωτηθείτε, άπαξ και υπάρχουν κάποια στοιχεία, πώς καταλήγουμε στα τελικά μας αποτελέσματα. Εδώ έχετε το προήμιο και εδώ έχετε ένα σύντομο έγγραφο, 25 σελίδες μόνο, όπου αναφέρονται οι διαδικασίες, οι κατευθυντήριες γραμμές που λένε ποιος κάνει την αξιολόγηση, πώς και σε ποιον δίνουμε τα αποτελέσματά μας, πώς συμμετέχουν οι διαφερόμενοι, ποια είναι τα επιστημονικά κριτήρια επίσης για την αναθεώρηση όσον αφορά τις επιπτώσεις στον άνθρωπο. Και αναφέρουμε επίσης και τη διαδικασία αποφάσεων. Τώρα, πέρα από το εξώφυλλο μέσα έχετε δύο κυρίως είδη πληροφοριών. Μπορείτε να πάτε και στην ιστοσελίδα μας και να τα διαβάσετε αν δεν βρίσκεται ενδιαφέρουσα την παρουσίασή μου. Εν πάση περιπτώσει, εγώ συνεχίζω. Θέλω να υπογραμμίσω εδώ κάποιες πτυχές στη διαδικασία μας που περιγράφονται ακριβώς μέσα στο προήμιο. Η, η ιεραρχία όσον αφορά την έρευνα για τον καρκίνο. Οι δικές μας οι μονογραφικές αξιολογήσεις βοήθησαν την ε, θεματολογία, την τερμινολογία, αλλά και καινοτομίες όσον αφορά τον εντοπισμό των ε, ερευνών και των αποτελεσμάτων. Διάφορες αξιολογήσεις μας έχουν ληφθεί υπόψη από κυβερνήσεις και από συστήματα αξιολόγησης κινδύνου σε διάφορες οργανώσεις και οργανισμούς. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ποιος κάνει τις αξιολογίες αυτές τις μονογραφικές από την οργάνωσή μας. Γίνονται από ανεξάρτητους επιστήμονες, εμπειρογνώμονες υψηλού επίπεδου που εμείς βρίσκουμε. Πρώτον, γιατί έχουν την πραγματογνωμοσύνη και δεύτερον, γιατί δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Όπως μπορείτε να φανταστείτε για τον κλήφοσετ αλλά και για άλλους καρκινογενείς παράγοντες υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι έχουν αξιόπιστους λόγους να βρίσκονται εκεί αλλά και κάτω από διαφορετικούς ρόλους ίσως. Γι' αυτό και εμείς εντοπίζουμε ότι μπορεί να είναι είτε πυρογνώμονες είτε αντιπρόσωποι ε, διεθνών ή εθνικών οργανισμών ή ως παρατηρητές από τη βιομηχανία ή από καθημαϊκούς ε, κύκλους ή και από την ίδια τη γραμματεία της οργάνωσής μας. Είμαι εγώ στη γραμματεία αυτή και βοηθούμε ώστε οι αξιολογήσεις να γίνονται με το σωστό τρόπο. Επίσης υπάρχει διαφάνεια κάθε φορά που υπάρχει σύγκρουση Ε, τα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας πριν από κάθε συνάντηση. Εδώ στην επόμενη διαφάνεια θέλω να σας εξηγήσω πώς σεβόμαστε την διαφάνεια. Πριν προχωρήσουμε σε μία αξιολόγηση υπάρχουν και στο προήμιο που είναι στην ιστοσελίδα μας, λέμε ποιο είναι το θέμα, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, ποιες είναι οι ομάδες εργασίας και ποιοι είναι αυτοί που συμμετέχουν. Τους αναφέρουμε πολύ πριν αρχίσει η διαδικασία. Είναι ανοιχτή η διαδικασία και σε επιστημονικούς παρατηρητές και ε, δημοσιεύεται στη συνέχεια και μπορεί κανείς να κατεβάσει τα αποτελέσματα δωρεάν. χρησιμοποιείται πολύ βιβλιογραφία. Τα έγγραφα υπάρχουν, μπορεί όποιος θέλει να τα συμβουλευτεί, να κρίνει και να λάβει υπόψη του όλους τους παράγοντες που λάβαμε και εμείς υπόψη μας για να προχωρήσουμε στην αξιολόγηση. Όλοι οι παράγοντες αναφέρονται και αναφέρονται ορθολογικά και τα αποτελέσματα. Τι είδους στοιχεία συμπεριλαμβάνουμε. Έχω μονογραφικές μελέτες που είναι πραγματικά πρωτότυπες. Ίσως να έχετε ακούσει τους όρους. Οι επιτροπές ε, συμβουλίων έχουν προτείνει τη συστηματική αναθεώρηση. Είναι κάτι το οποίο ε, θεωρούν ότι βοηθάει. Και έτσι χρησιμοποιούμε και εμείς μία δομή ιεραρχικής αξιολόγησης η οποία μας, μας βοηθάει στη δουλειά μας. Πρόκειται λοιπόν για μια ιεραρχική δομή. Σε αυτή τη διαδικασία τώρα κάθε μελέτη αναθεωρείται, είτε έχουμε θετικά είτε αρνητικά αποτελέσματα, αξιολογούμε τα δυνατά και τα δύνατα σημεία της κάθε μελέτης. Η ομάδα εργασίας χρησιμοποιεί και αγγίλες για να περιγράψει, να βάλει σχόλια τα οποία βοηθούν να καταλάβει κανείς γιατί κατέληξαν στην αξιολόγηση που κατέληξαν. Υπάρχουν λοιπόν όλες οι πληροφορίες. Επόμενη διαφάνεια. Πώς όλα αυτά συγκεντρώνονται τώρα και προχωρούν στο χρόνο. Πορτοκαλί. Βλέπετε τι κάνει η γραμματεία των μονογραφικών προγραμμάτων. Συντονίζει όλες τις πλευρές ε, της συνάντησης. Μετά έχουμε τα μέλη της ομάδας εργασίας 8 μήνες πριν τη συνάντηση κάνουν την μελέτη, αξιολόγηση, βάζουν τα σχόλιά τους σε αγγείλες και ενημερώνουν τους ομολόγους τους. Και στη συνέχεια γίνεται η συνάντηση. Πρώτα απ' όλα ανακοινώνουμε τους συμμετέχοντες και τις άλλες κατηγορίες επιστημόνων. Και μετά έρχεται το προσωπικό στη Εκεί γίνονται συναντήσεις με τους επιστήμονες και εκεί καταλήγουμε στα συμπεράσματα. Μετά υπάρχει μια σύντομη δημοσίευση με την, ε, που ονομάζεται The Lancet Oncology Publication και στη συνέχεια μοιραζόμαστε τα αποτελέσματά μας με διάφορες οργανώσεις υγείας και τέλος δημοσιεύεται η μονογραφική μελέτη για τον Glyphosat, για παράδειγμα, έγινε τον Ιούλιο του 2015. Η χρονιά ήταν ε, πολύ γεμάτη για μας. Για τον Glyphosat τώρα, πιο συγκεκριμένα. Να τι περιλαμβάνει η μονογραφική μας μελέτη. Πάντα υπάρχουν οι γενικές παρατηρήσεις και μετά υπάρχει αυτό που λέμε η κριτική αναθεώρηση των δεδομένων. Θα επικεντρωθώ εδώ στον καρκίνο, στους ανθρώπους, στα ζώα και την ε, μηχανιστική και άλλα δεδομένα. Στη συνέχεια η αξιολόγηση αναφέρεται στα δύο τελευταία τμήματα της μονογραφικής μελέτης. Και υπάρχουν βέβαια και τα σημεία αναφοράς. Πώς γίνεται λοιπόν η μονογραφική αξιολόγηση. Υπάρχουν τριών ειδών στοιχεία. Υπάρχει συστηματική μελέτη και εδώ βλέπετε την ορολογία που χρησιμοποιούμε. για τα καρκινογενή, για τους ανθρώπους και για τα ζώα. Τα στοιχεία τα καθορίζουμε σε κατηγορίες. Αν υπάρχουν επαρκή αποδυτικά στοιχεία, περιορισμένα στοιχεία, ακατάλληλα ή κάποια τα οποία δείχνουν ότι δεν πρόκειται για καρκινογενή παράγοντες είναι μεθοδολογία που χρησιμοποιούν και άλλες αξιολογήσεις. Στα μηχανιστικά και άλλα σχετικά στοιχεία υπάρχει το αδύναμο, το μέτριο, το ισχυρό αποδεικτικό στοιχείο. Και όλα αυτά τα χρησιμοποιούμε στη συνολική αξιολόγηση. Και εδώ βλέπετε τις ομάδες που σας περιέγραψα και στην αρχή, 1, 2α, 2β κλπ. Τώρα τα στοιχεία για τον γλυφοσάτ. Θα σας εξηγήσω πώς τα συμπεριλάβαμε στην συστηματική μας προσέγγιση. Οι επιδημιολογικές ε, μελέτες συμπεριλαμβάνουν μελέτες που έχουν γίνει από τον non-Hodgkin λιμφώμα. Όπως επίσης από μελέτες που έχουν από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Σουηδία. Έχουμε μελετήσει και άλλα παρασιτοκτόνα. Επίση, έχει γίνει μια άλλη μεγάλη γεωργική μελέτη στι ΗΠΑ που δεν πρόσθεσε όμω στοιχείο. Συνολικά, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι έχουμε ε, περιορισμένες αποδείξει για το κατά πόσο πρόκειται για καρκινογενή παράγοντα όσον αφορά τους ανθρώπους. Λέμε όμως ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η περίπτωση του να είναι όντω καρκινογενή. Μελετήσαμε ασενικά ποντίκια σε μεγάλο αριθμό. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι σε δύο μελέτες με ποντίκια διαπιστώθηκε ε, συσχετισμός με όγκους που παρατηρήθηκαν στα ποντίκια αυτά. Και στις δύο μελέτες λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχουν πιθανότητες για συσχετισμό με την ουσία. Βάση δύο ανεξάρτητων μελετών. Τέλος, τις μηχανιστικούς παράγοντες. Έχουν γίνει εκατοντάδες μελέτες. Εμείς τις ταξινομήσαμε σε δέκα κατηγορίες και καταλήγουμε ότι σε δύο περιπτώσεις έχουμε ισχυρές ενδείξεις για τοξική επίδραση στα γονίδια, για παράδειγμα, και λέμε ότι πρόκειται για παράγοντες που όντως μπορεί να οδηγούν σε καρκίνο. Εδώ θα σας δείξω πώς καταλήξαμε στην αξιολόγηση της ομάδας 2α για καρκίνο σε ανθρώπους. Είπαμε ότι έχουμε περιορισμένα στοιχεία. Σε περίπτωση καρκίνου στα ζώα επαρκής αποδείξεις, ότι δηλαδή κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να είναι καρκινογενή αρκές στους ανθρώπους και υπάρχουν και τα μηχανιστικά στοιχεία που λένε ότι βάσει πειραμάτων που γίνονται στα ζώα έχουμε ισχυρές ενδείξεις. Η αξιολόγηση αυτή λοιπόν για το γλυφοσάτ που είναι το θέμα σήμερα έχει γίνει και για άλλους παράγοντες, για άλλες ουσίες με διαφορετικά επίπεδα στοιχείων. Είχαμε ταξινόμηση 2β σε δύο περιπτώσεις και δύο άλλες περιπτώσεις 2α. Συνοπτικά, ελπίζω να σας περιέγραψα ότι ανεξάρτητα ε, γίνονται οι μελέτες αυτές και ότι γίνεται συστηματική αξιολόγηση και αναθεώρηση. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you very much. And now we give uh, immediately the floor to the EFSA expert. Και τώρα περάσουμε στον πρόσωπο της EFSA. Thank you very much, Mr. Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Αποτελεί χαρά πάντα για μας να ερχόμαστε στο Κοινοβούλιο και να συζητάμε το πλαίσιο και το υπόβαθρο των ε, μελετών της ΕΦΣΑ. Θα ήθελα να προτού να σας αναφέρω τα συμπεράσματα της μελέτης, να σας μιλήσω για το πλαίσιο της εργασίας μας σχετικά με το glyphosate. Έχουμε μια διαδικασία τριών ε, βημάτων προτού να εγκριθεί ένα προϊόν σε μια ένα Το πρώτο βρισκόμαστε στο πρώτο βήμα, το pre-market ή την αξιολόγηση κινδύνου η την αξιολογηση κινδυνου μια ουσια και μετα γινεται από τα 28 κράτη-μέλη. Εργαζόμαστε εδώ με 600 εμπειρογνώμονες σε ένα δίκτυο και ασχολούμεθα με τον τομέα των φυτοφαρμάκων στα 28 κράτη-μέλη. Μετά από το το πρώτο αυτό βήμα η Ευρωπαϊκή Κομισιόν λαμβάνει απόφαση για την έγκριση ή μη έγκριση αυτής της ουσίας και μετά πέραμε στο τρίτο φάση όπου η αξιολόγηση κινδύνου γίνεται αυτή τη ουσία στην γεωργία ή αλλαχού. Τώρα βρισκόμαστε στο τριτο φαση οπου η εξολογηση κινδυνου γινεται για καθε προιον που χρησιμοποιειται στην γεωργια η Ελλακού. τωρα βρισκομαστε στο σταδιο 1. Επόμενη διαφάνεια. Αυτό το οποίο κάναμε εδώ είναι μια συντολική αξιολόγηση κράτησε τρία χρόνια, ξεκίνησε το 2012 με την ε, Γερμανία ως ε, εισηγήτρια και κάναμε αυτή την ε, peer review με τους εμπειρογνώμους από τα 28 κράτη-μέλη. Υπήρχαν περίπου 100 εμπειρογνώμονες οι οποίοι συμμετείχαν στην εργασία της peer review και Φυσικά χρησιμοποίησαν, ε, χρησιμοποίησαν όλα τα διάφορα Ινστιτούτα και οργανισμούς που είχαν, ε, ε, είχαν ήταν εγκεκριμένα από τα κρατημέλη. Και υπήρχε επίση και ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, συμμετείχε και από τι ΗΠΑ η ΕΠΑ. Ε, ε, διαδικασία διαφανής διότι κάναμε μια δημόσια διαβούλευση στην αξιολόγηση που έκανε η Γερμανία. Φυσικά δημοσιεύτηκε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης και όχι μόνο δημοσιεύσαμε τα συμπεράσματα αλλά και όλα τα έγγραφα που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας περίπου 6.000 σελίδες έγγραφα τα οποία περιλαμβάνουν ακόμα και τα σχόλια και αποτελούν το υπόβαθρο των όσων χρησιμοποιήσαμε και αξιολογήσαμε. Συμπεριλαμβανομένων επίση και τι μελέτε των βιομηχανιών. Το, το σύνολο των ε, πληροφοριών που έχει δημοσιεύσει η ΕΦΣΔΑ είναι κάτι το οποίο θα το βρείτε στην επιστημονική ε, βιογραφία και ο ΠΟ έχει ζητήσει τα σχετικά στοιχεία για την αξιολόγηση η οποία είναι στα σκαριά. Τώρα θα δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου που θα σας ε, παρουσιάσει τα βασικά συμπεράσματα αυτής της ε, peer review. Ευχαριστώ Μπέρναρτ. είχαμε μια συνολική αξιολόγηση των ε, τοξικολογικών και μη δεδομένων. Καλύψαμε το όλο πλαίσιο των ε, πληροφοριών με την, για την τοξικότητα το ε, βασιστήκαμε πάνω στις σύγχρονες μελέτες που έχουν γίνει και προτείνουμε κάποιες νέες αξίες τοξικολογικές οι οποίε θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση κατά τη διάρκεια έκθεσης ε, σε αυτήν την ουσία. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι είναι η πρώτη φορά που έχει προταθεί μια τέτοια διαδικασία για το γλυφοσάιτ σχετικά με την αξιολόγηση της ε, καρκινογένειας ε, όταν με και άλλες ε, υπηρεσίες, ε, ακολουθούσαμε την διαδικασία του ARK. Κάναμε την αξιολόγηση που ακολουθούσαμε μάλλον αξιολόγηση που έκανε η Γερμανία σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη βασιζόμενοι στα κριτήρια της κανονισμού CLP που συμφωνήθηκε μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για την αξιολόγηση των χημικών ουσιών. Κάναμε λοιπόν την αξιολόγηση της, του γλυφοσέιτ. Ο κανονισμός CLP βασίζεται στο εναρμονισμένο σύστημα το οποίο ε, έχει αναπτύξει ΙΕ, ιδιαίτερα για την ταξινόμηση των χημικών ουσιών. Και όπως ε, υπόθηκε ήδη η IRC ακολουθεί με διαφορετική ταξινόμηση τα δύο στοιχεία που ήταν, παίζαν ρόλο όταν ξεκίνησε η μελέτη ήταν πρώτον να διασφαλίσουμε ότι καλύπτουμε όλα, όλες τις ε, φυστάμενες μελέτες διότι στο πλαίσιο των μονογραφιών λάβαμε υπόψη διάφορες επιδημιολογικές μελέτες και ελέξαμε όλες τις αναφορές που προέκυψαν από νέε μελέτες. Το δεύτερο στοιχείο ήταν να έχουμε μια πλήρη αξιολόγηση επιστημονικής φύσης ε, ακολούσαμε ακριβώς τους ίδιους ε, κανόνες που ε, εφάρμοσε και η ΕΦΣΑ βασιζόμενες σε επιστημονικά στοιχεία και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για μας. Κάναμε μια αξιολόγηση για το θέμα της καρκινογίας. Γένειας και στο οποίο συμπερίληψαν 30 εμπειρογνώμονες της ΕΦΣΑ αλλά και από οργανισμούς ε, από άλλους οργανισμούς ευρωπαϊκούς και επίσης από τον ε, ΠΟΕ και από την UPSA οι οποίοι συμμετείχαν ως παρατηρητές της συζήτησης μας για την αξιολόγηση των ανθρώπινων επιδημιολογικών δεδομένων έχουμε ακριβώ τι ίδιε πληροφορίε που η IARC παρουσίασε στην μονογραφή. Και εφαρμόζαμε τα κριτήρια του CLP και τα συμπεράσματα είναι ότι υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία για την, για την καρκίνου στον άνθρωπο για τις ε, μελέτες ε, επί των ζώων έχουμε πολλές, πολύ περισσότερα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην αξιολόγηση. Έχουμε 13 ε, μελέτες για τα για τα μυρικαστικά. Όλες τις μελέτες ελέγχθησαν προσεκτικά από τους επιστήμονες της ΕΦΣΑ και τα κράτη-μέλη και υπήρξαν ε, ε, αποδείξεις σύμφωνα με τον κονισμό CLP ότι οι κατελτές γραμμές ε, είναι σύμφωνες με αυτή της, των συστάσεων της, του ΟΣΑ. Το μηχανιστικός, μηχανιστική προσέγγιση που παρουσίασε η ΑΕΡΚ είναι ότι το γλυφοσέτ δεν είναι ιδιαίτερα τοξικό και αυτό και έχουμε 13 μελέτες οι οποίες αναφέρουν αρνητικές επιπτώσεις ε, έχουμε λίγες μελέτες, τρεις συγκεκριμένα που προτείνουν ότι παρέχουν κάποια τοξικότητα. Ε, αυτές οι μελέτες ε, ελέγχθηκαν προσεκτικά και τα συμπεράσματα είναι ότι η τοξικότητα είναι χαμηλή και άρα δεν θα πρέπει να ταξινομηθούν σχετικά με την τοξικότητα του glycoside. Όχι, όχι για το γλυφοσέτ, αλλά για, για άλλα προϊόντα είχαν θετικές επιπτώσει. Υπάρχουν και άλλες μελέτες λοιπόν, οι οποίες αναφέρουν αρνητικά αποτελέσματα και υπάρχουν αρκετά συμπεράσματα στι μονογραφίε, που δείχνουν αρνητικές επιπτώσει. Παζόμενα λοιπόν σε αυτά τα αποτελέσματα, στα συμπεράσματα, συστήνουμε τα κράτη-μέλη να έχουν ιδιαίτερη, να προσέξουν ιδιαίτερα το θέμα της τοξικότητας ε, κατά την έγκριση για την ε, πρόθεση στην αγορά των προϊόντων. Uh, uh, Για την καρκινογέννηση έχουμε κάποιες μελέτες ε, μεταξύ αυτών κάποιες είναι θετικές ε, και αρνητικές ανάλογα με την ε, στατιστική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται. Η ΕΦΣΑ προτιμάει την μεθοδολογία που συμπεριλαμβάνεται στην μελέτη του ΟΖΑ. Άλλοι χρησιμοποιούν διαφορετική προσέγγιση, αξιολογούν τα δεδομένα και με βάση τα, τα, τα αποτελέσματα κάνουν την κατάλληλη αξιολόγηση. Για την ΕΦΣΑ, η βιολογική σημασία των ε, μελετών ε, σχετικά με την καρκινογέννηση στους ανθρώπους θεωρούν ότι είναι ιδιαίτερα χαμηλή δεν διαπιστώσαμε ότι υπάρχει α, ασυμφωνία ανάμεσα στις δύο μελέτες Υπάρχει υψηλή τοξικότητα που δεν συνδέεται με την καρκινογέννηση και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί λοιπόν ως ε, αξιόλογο στοιχείο για την ε, χαρακτηρισμό ως καρκινογενή. ECD των, ε, των αποτελεσμάτων. Κάναμε, συγκρίναμε όλες τις μελέτες και ανάλογα με τα κριτήρια αξιολόγηση της, CLP θεωρήσαμε ότι το glyphosate ε, δεν, ε, είναι δεν προκαλεί καρκινογέννηση. 27 κράτη-μέλη της Ένωσης στηρίζουν την έψη σε αυτή την αξιολόγησή της. Υπάρχει μια άποψη τη ε, της Σουηδίας η οποία αφορά το ζήτημα και ως αυτού του θεωρεί ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην κατηγορία 2 σύμφωνα με τη CLP. Αυτά που προτείνουν τα αποτέλεσματα της ε, ΕΦΣΑ είναι ότι δεν θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις ε, καρκινογόνες ουσίες ε, και ακόμα αν ε, ληφθεί υπόψη η άποψη για τη συμβίωση στην κατηγορία 2. Συμπερασματικά κάνω μια συνολική επιστημονική αξιολόγηση χρησιμοποιώντα υψηλότερα ε, αποδεικτικά στοιχεία από την ΙΑΡΚ. Η αξιολόγηση έγινε σύμφωνα με τον κανονισμό που αποφάσισε το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο 1007 του 2007. Αυτέ οι προφορίε θα συμπληθούν από την Κομισιόν στην σχετική διαδικασία και από τα κράτη-μέλη στην αξιολόγηση. Εξετάσαμε επίση το ζήτημα τη ε, καρκινογέννηση εφαρμόζοντα τα κριτήρια σύμφωνα με το ΣΕΛΠ, θεωρούμε ότι το βλέφο δεν θα πρέπει να ταξινομηθεί ως κακινογόν ουσία. Όπως ήδη ανέφερα, 27 κράτη-μέλη στηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Υπάρχει μια άποψη της μειοψηφία για την συμπερίληψη την κατηγορία 2 της ουσίας και δεν υπάρχουν άλλα κράτη που να υποστηρίζουν την συμπερίληψή τους στην κατηγορία 1. Η αξιολόγηση έχει αναφερθεί, όπως είπε και ο Μπέρναρτ, έχουμε δημοσίευσει πάνω από 6.000 σελίδες με όλες τις λεπτομέρειες κάθε επιμέρους μελέτης που έγινε και απαντήσαμε σε όλα τα σχόλια στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης. Επιπλέον, σύμφωνα με την ε, ορισμό CLP, Νομίζουμε ότι διατηρήσαμε την ε, σωστή εφαρμογή του κανονισμού. Ευχαριστώ λοιπόν κύριε Πρόεδρε για την δυνατότητα που μας δώσατε να ε, κάνουμε αυτές τις δηλώσεις σήμερα και είμαστε στη διάθεση για κάθε διαφορετική. Ευχαριστώ. δεν ξέρω αν υπάρχουν ε, ερωτήσεις από τους ευρωβουλευτές. Υπάρχουν ο κύριος Πέτερλε από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν περίμενα να είμαι ο πρώτος, λέει ο κύριος Πέτερλε. Θέλω να σας πω ότι είμαι ευγνώμων για αυτές τις ε, δύο που ακούσαμε. Νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμες αυτές οι επιστημονικές μελέτες γιατί και οι δύο καταλήγουν το συμπέρασμα ότι η αξιολόγηση ε, θα πρέπει να γίνεται με περιεκτικό και ανεξάρτητο τρόπο. Για μας λοιπόν είναι σημαντικό να μπορούμε να κατανοήσουμε τη διαφορά. Γιατί <clears throat> στη μία περίπτωση αναφέρεται ότι το γλυφοσάτ κρίνεται ως καρκινογενές ε, σε ανθρώπινα όντα. Η δεύτερη μελέτη καταλήγει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Και παρακολούθησα, άκουσα πολύ προσεκτικά αυτά που είπε η ΕΦΣΑ. Επίσης ε, η ΕΦΣΑ ανέφερε ότι υπάρχουν κάποια ε, στοιχεία σε σχέση με τον κλειφωσάτ που πρέπει να διευκρινιστούν περαιτέρω. Και εγώ θεωρώ ότι θα ήταν καλύτερα να μην αποφασίσουμε πριν τελικά δοθούν αυτές οι περαιτέρω διευκρινήσεις γιατί νομίζω ότι ε, οι αξιολογήσεις αφορούν και το καθαρό γλυκοσάτ και το άλλο παράγωγα ίσως του γλυφοσάτ. Αυτό νομίζω ότι είναι καθοριστική σημασία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα το οποίο μας απασχολεί, το γλυφοσάτ. <coughs> Έχουμε δώσει παράταση για να έχουμε περισσότερο χρόνο, για να ε, αντιμετωπιστεί για να υπάρξει την μελέτη. Και σήμερα έχουμε τους δύο αρμόδιους οργανισμούς, τον ΙΑΡΚ και την ΕΦΣΑ. Και ρωτώ τον ΙΑΡΚ, στη μελέτη σας, τον γλυφοσάτ, συγκρίθηκε με άλλες ουσίες. Εξετάστηκαν άλλες ενώσεις ουσιών. Αυτή ήταν η ερώτηση προς την ΙΑΡΚ και η άλλη προς την ΕΨΑ. Στη μελέτη της ΕΨΑ, γιατί δεν εμφανίζεται το γλυφοσάτ ότι υπάρχουν ε, ε, διευμοί ως προς το προϊόν αυτό. Ε, δεν αναφέρεται τίποτα στη μελέτη σας και αυτό με εκπλήσει και ίσως μπορείτε να μας πείτε πώς είναι δυνατόν να μην έχετε μελετήσει αυτά τα συγκεκριμένα θέματα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε η κυρία Χάζενκαμπ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο τρόπος με τον οποίο δίνεται η γνωμοδότηση για το γλυφοσάτ είναι σκανδαλώδης. Το γλυφοσάτ κινδυνεύει να γίνει το σύμβολο του τι δεν πάει καλά στην Ευρώπη. Η γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ λοιπόν για το γλυφοσάτ βασίζεται σε έρευνες, λέει περισσότερες από εκείνες του ΙΑΡΚ, αλλά οι πηγές δεν δημοσιεύονται. Δεν υπάρχει διαφάνεια. Και βασίζεται κυρίως στο Γερμανικό Ινστιτούτο για την Αξιολόγηση Κινδύνου. Είναι σκανδαλώδες. Εμείς οι Ολλανδοί συνάδελφοι θέλουμε την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα όταν πρόκειται για τα τρόφιμά μας. Η ΆΡΚ έκανε πάρα πολλές μελέτες και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το γλυφοσάτ είναι πιθανώς καρκινογενές. Πρόεδρε, υπάρχει και επιστολή επιστημόνων που καταδικάζουν την έλλειψη διαφάνεια στην ΕΦΣΑ. Έτσι λοιπόν κάνω και εγώ έκκληση για να ζητήσω το γλυφοσάτ να μην επιτρέπεται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να κάνει περισσότερα για να αποφύγει την χρήση του και οι άλλες ομάδες το ίδιο νομίζω ότι θα στήσουν από την Επιτροπή. Και αν δεν βρίσκετε λόγους για να απαγορεύσετε απευθείας μέχρι τώρα το γλυφασάτ, τώρα νομίζω έχετε λόγους και μπορείτε να το κάνετε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κυρία Γκέρλινγκ. Τζούλη, έχεις το λόγο. αν νόμιζα ότι ήμουν τελευταία, αλλά όχι από ό,τι φαίνεται. Θέλω να ρωτήσω κάτι δεν αναφέρομαι στην ίδια επιστολή των επιστημόνων, αλλά κάποιες πληροφορίες που αναφέρονται εκεί. Φαίνεται ότι υπάρχει διαμάχη ανάμεσα στην BFR και την ΙΑΡΚΑ e όσον αφορά τα στοιχεία που χρησιμοποιούν Όσοι υπέγραψαν την επιστολή αυτή υποστηρίζουν ότι στην αξιολόγηση της ΕΦΣΑ υπήρχαν ε, αρκετά βάσιμα δεδομένα που έδειχναν ότι δεν ήταν ε, κάτι με διαφάνεια, ότι δεν υπήρχε αξιοπιστία τελικά. Και έχουμε να κάνουμε με καρκινογέννηση, έτσι. Οπότε λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω την ΕΦΣΑ, όντως είναι έτσι συμπεριέλαβαν στοιχεία στην αξιολόγησή τους που δεν είναι διαθέσιμα σε κανέναν άλλον, ούτε στην ΙΑΡΚΑ, ούτε σε άλλους ε, όπως καταγγέλουν οι επιστήμονες. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Εκάιτ. Α, η κυρία Διβάζη πρώτα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Έχω πολλές ερωτήσεις για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτον, είναι αλήθεια ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε για το γλυφοσάτ να υπάρξει μια σχέση αιτία του ισχυρή και όχι sufficient evidence όσον αφορά την χρήση του γλυφοσάτ και την παρουσία καρκινογένεσης. Δεύτερη ερώτηση προς την ΕΦΣΑ και το και η κυρία Γκέρλινγκ. Πράγματι, ακούμε ότι το BFR ε, χρησιμοποίησε μελέτες αναφοράς ε, για την ε, τοξικότητα του γλυφοσάτ που δεν δημοσιεύτηκαν μετά. Και μετά μαθαίνουμε ότι ένα τρίτο των εμπειρογνωμόνων για τα παρασιτοκτόνα ουσιαστικά δουλεύουν στον αγροτικό τομέα και χρηματοδοτούνται από εκεί. Τέλος, το πιο σημαντικό, το γλυφοσάτ είναι μια ενεργός ουσία δραστήρια. Όταν τη χρησιμοποιούμε χρησιμοποιούμε είναι τα, οι ουσίες οι οποίες δημιουργούνται από την χρήση που έχουν σαν αποτέλεσμα ταξικότητα να είναι πολύ μεγάλη. Αυτό λοιπόν που θέλω να ρωτήσω είναι η Μονσάντο που κάνει αυτές τις μελέτες είναι αλήθεια ότι δεν δίνει ε, τα στοιχεία για τα προσθετικά τα οποία χρησιμοποιεί. Είναι αλήθεια ότι όταν κάνει την αξιολόγησή της η ΕΦΣΑ χρησιμοποιεί μόνο τον γλυφοσάτ και όχι το Roundup με όλα αυτά τα πρόσθετα τα οποία είναι, πολύ τοξικά. Πήγαμε στην Πάρμα, βρεθήκαμε με την άφησα, τους είχαμε πει προσοχή, το Ιάρκα κάνει μια αξιολόγηση και εσύ προσοχή γιατί θα την πατήσετε. Και τελικά για άλλη μια φορά κάνατε το ίδιο λάθος, κάνατε μια αξιολόγηση η οποία λαμβάνει υπόψη ένα μικρό μέρος των στοιχείων και δεν συμπεριλαμβάνει και το ραντόπ που είναι πολύ τοξικό. 96 εμπειρογνώμονες ε, λοιπόν ζήτησαν ε, το λογαριασμό από την ΕΦΣΑ και είπε γιατί είπαν γιατί υπάρχει τόσο διαφορετική αξιολόγηση από την ΕΦΣΑ και από την ΕΑΤΚΑ. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι προς τιμή σας όλα αυτά, αν μη τι άλλο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Άκουσα όπω και όλοι οι υπόλοιποι πολύ προσεκτικά τη συζήτηση, βρίσκω ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, αλλά θα ήθελα να πάω στη θέση των πολιτών. Διότι υπάρχει το ΙΑΡΚ, το Κέντρο για την Έρευνα του είναι η Διεθνή Οργάνωση για την Υγεία και είναι και η ΕΦΣΑ. Και στην πρώτη περίπτωση έγιναν μελέτε για τα προϊόντα τα οποία είναι στο, τυχάνουν εμπορίας με αποτελέσματα ε, ότι τα αποτελέσματα ήταν ανεπαρκή για το θέμα της, ε, του καρκίνου, που προκαλούν καρκίνο στον άνθρωπο. Υπήρξαν λοιπόν αποτελέσματα από, και από άλλη εταιρεία, την υπηρεσία την ΕΨΑ, ότι δεν υπάρχουν τέτοιες ανθρωπιστικά στοιχεία. Αφενός ε, έγινε κριτική για την συμπερίληψη στοιχείων που περιλαμβάνουν τα πειράματα σε ζώα, αλλά αυτή είναι η προσέγγιση η οποία γίνεται στον επιστημονικό κόσμο γενικά, τώρα στον τομέα τη υγείας. Δεν καταλαβαίνουν λοιπόν γιατί τώρα τίθεται να αμφιβόλο αυτή, σε αυτή την περίπτωση. Αλλά μια διαδικασία διάφανη και στην δεύτερη περίπτωση, το Γερμανικό Ινστιτούτο για να Αξιολόγηση του Κινδύνου ε, και η ΕΦΣΑ δεν ε, έδωσαν ε, και δημοσίευσαν τα στοιχεία για την, υποστήριξη, για την θέμα του βιομηχανικού απορρίτου. Άρα λοιπόν κρυβόμαστε πίσω από το βιομηχανικό απόρριτο για τα θέματα υγείας. Η Επιτροπή αναφέρεται σε μια ε, συζήτηση εμπειρογνωμόνων στην οποία συμμετέχουν διάφοροι εμπειρογνώμονες εταιριών όπως η Bayer. Ε, και τελειώνω, κλείνω να πω τα Η ΕΦΣΑ ε, κάνει μια προσέγγιση, λέει στατιστική, από στατιστική σκοπιά, δεν υπάρχουν σίγουρα αποτελέσματα αλλά δεν βρισκόμαστε ακριβώς στην περίπτωση για την εφαρμογή της ε, αρχής της πρόληψης. Ευχαριστώ Πετιτσίνη. Το κράδενα το σφυράκι απλά για τον χρόνο, για κανένα λόγο. Η κυρία Γιωτό. Ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να πω ότι άκουσα τις ε, μελέτες σε κάθε επιστημονική μελέτη το πρώτο που έχει σημασία είναι το υλικό και η μεθοδολογία. Για τα δύο αυτά δεν συμφωνούν μεταξύ τους η ΕΦΣΑ και η ΑΡΚΟ, οπότε δεν μου κάνει εντύπωση που τα αποτελέσματα είναι διαφορετικά. Η ΕΦΣΑ, από ό,τι φαίνεται, έχει δουλέψει με την ενεργό ουσία, ενώ οι άλλοι χρησιμοποίησαν τον πλήρη τύπο με τα βοηθήματα, τα βοηθητικά. Θα πρέπει όμω να διευκρινιστεί αυτό. Για το γλυφοσάτ υπάρχουν 30 εμπορικά προϊόντα και το καθένα από αυτά σίγουρα χρησιμοποιεί διαφορετικά adjuvant βοηθητικά. Και υπάρχει και μία άλλη μελέτη της κοινή Επιτροπής ε, Φυτοφαρμάκων του ΠΟΕΤ, Παγκόσμιας Οργάνωσης ε, Υγείας, του ΠΟΕΤ, που έχει τα ίδια αποτελέσματα με την ΕΦΣΑ. Εμείς που δεν είμαστε πυρογνώμονες για το θέμα αυτό, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά μας δημιουργούν σύγχυση και πολλοί θα θέλαμε να διευκρινιστούν οι μελέτες, να χρησιμοποιούν τα ίδια υλικά, την ίδια μεθοδολογία και τα ίδια βοηθητικά. Υπάρχουν 30 διαφορετικοί χημικοί τύποι για τη χρήση του γλυφοσάτ. Και θα ήθελα και σχόλια περισσότερα για την επιστολή αυτή που εστάλει στην Επιτροπή από τους επιστήμονες κλπ. Ευχαριστούμε. Κύριε Σπότς. Θα ήθελα να είμαι σύντομος, πολύ σύντομος. Ε, κοιτάξτε, και εγώ το κοίταξα λιγάκι το υλικό και η μεγαλύτερη διαφορά δεν έγκυται στο ότι η μία πλευρά δούλεψε μόνο με την ουσία και οι άλλοι με τους κινδύνους. Ε, εγώ νομίζω ότι ο μεγαλύτερος, ε, κινδυ... μεγαλύτερη διαφορά, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι μία πλευρά ε, χρηματοδοτήθηκε από τη βιομηχανία. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε αυτό. Εγώ θέλω να ρωτήσω, γιατί προβλέπετε αδειοδότηση για 15 χρόνια, τη στιγμή μάλιστα που επικρατεί μεγάλη ασάφεια. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Εάν η Επιτροπή επιτρέψει, δώσει άδεια για αυτό το προϊόν για το μέγιστο χρονικό διάστημα που επιτρέπεται, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Σας είπα, τη στιγμή που δεν είμαστε καν σίγουροι. Στους ε, ενδοκρινικούς ε, καταστροφείς ε, εκεί, γιατί δεν προβλέπεται αναθεώρηση, Επίσης ε, με ενδιαφέρει εκεί που γίνεται λόγος για το ότι το γλυφο, γλυκοσάτ επηρεάζει πολύ σοβαρά τα ένζημα 85, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πάρα πολλές ασθένειες, συμπεριλαμβανομένου και του καρκίνου και ε, δεν το κατανοώ γιατί δεν αναφέρεται αυτή η μελέτη. Πρόκειται για μια ε, ιδιαίτερα περιεκτική αμερικανική μελέτη η οποία ε, περιγράφει αυτό το πρόβλημα. Και θέλω να σας πω το εξής. Για μας, για τους ευρωβουλευτές, αυτή η κατάσταση είναι παντελώς απαράδεκτη. γιατί νομίζω ότι πρέπει να εφαρμόζουμε την αρχή της πρόληψης. Κοιτάξτε κύριε Πρόεδρε, πράγματι υπάρχουν επιστημονικές μελέτες που δείχνουν ότι το φυτοφάρμακο γλυφοσάτ συνεπάγεται κινδύνους ε, για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων και ενδέχεται να οδηγήσουν και σε εμφάνιση καρκίνου. Μπάση τόση δεν αποκλείεται αυτό. Άρα δηλαδή είναι επισημάνσεις ε, οι οποίες δικαιολογημένα ε, οδηγούν στο να έχουμε αμφιβολίες για αυτό το φυτοφάρμακο. Άρα δηλαδή εδώ ισχύει η αρχή της πρόληψης. Το γλυφοσάτ και όλα τα προϊόντα που περιλαμβάνουν γλυφοσάτ οφείλουν να αποσυρθούν από την αγορά. Και είναι ντροπή ορισμένες πολιτικές ε, ομάδες ε, να μην... Μισό λεπτό διακόπτει ο πρόεδρος. Υπήρχε κάποιο πρόβλημα με την αγγλική μετάφραση, τώρα λύθηκε. Λοιπόν, μπορείτε να συνεχίσετε. Τώρα να τα πω από την αρχή. Όχι, όχι, εντάξει, πέστε τα από εκεί που είχατε σταματήσει. Λοιπόν, ε, θα ήταν σκάνδαλο μία μειοψηφία ε, της Επιτροπής Ενδύει να μπλοκάρει την Επιτροπή των Πρασίνων που είναι να αποσυρθεί τον Γλυφοζάτ. Ε, θα ήταν απαράδεκτο αυτοί οι συνάδελφοι να προσκυνήσουν οικονομικούς παράγοντες αντί να λειτουργήσουν προληπτικά για τον άνθρωπο και για τα ζώα. Απευθύνομαι στη συνείδησή σας να μην συμβάλλετε το να γίνονται παιχνίδια, επιπόλαια παιχνίδια με την υγεία των ανθρώπων στην Ευρώπη. Γιατί αλλιώς σας είπα θα γίνουμε οι προσκυνητές των πολυεθνικών. Ähm, es ist wie gesagt worden, Κοιτάξτε, στη Γερμανία σε 40% των εκτάσεων χρησιμοποιείται το γλυφοσάτ. Δηλαδή υπάρχει αυτό. Ε, δεν μπορούμε να το απαρνιόμαστε. Και όχι γιατί το χρειάζονται οι άνθρωποι, αλλά και γιατί είναι και φτηνό, να το πούμε και αυτό. Υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις που είναι πιο ακριβές. Αυτό που με εκπλήσει στη γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ είναι ότι έχουν αυξήσει τη μέγιστη δυνατή πρόσληψη σε μερίσια βάση από το 0,3 στο 0,5. Και αυτό δεν εξετάζεται ούτε το ότι το ε, γλυφοζάτ χρησιμοποιείται και λίγο πριν από τη συγκομιδή. Και αυτό είναι αυξημένος κίνδυνος. Θα ήθελα να μάθω την ε, θέση ε, στην επιστολή 96 επιστημόνων που σας ε, κατηγορούν ότι δεν εφαρμόζετε την οδηγία 96 του ΩΣΑ. Είναι πολύ αυστηρή και σκληρή αυτή η κατηγορία. Πρέπει λοιπόν να τοποθετηθείτε από αυτού. Εδώ με συγχωρείτε πρόκειται για την αξιοπιστία της πολιτικής μας και κατά πόσον προστατεύουμε τον πολίτη όχι. Γιατί αν υπάρχει κίνδυνος ε, δεν είναι δυνατόν λέμε υπάρχουν διαφορετικέ αξιολογίε. Όχι, στι περιπτώσει αυτέ είμαστε αναγκασμένοι να εφαρμόζουμε την αρχή τη πρόληψη και δεν καταλαβαίνω πώ είναι δυνατόν η ΕΦΣΑ. Παρότι είχε έξι μήνε, η ΕΦΣΑ έτρεξε να υιοθετήσει τη μελέτη του Γερμανικού Ινστιτούτου Αξιολόγηση Κινδύνων χωρί να επεξεργαστεί τη μελέτη της ΙΑΡΚ. Ε, ναι μεν είναι θέμα των ε, κρατών μελών, αλλά είναι και θέμα το ότι ε, δεν μπορεί κανείς ε, την αξιολόγηση να την παραπέμπει στα κράτη-μέλη. Δεν είναι δυνατόν η ΕΦΣΑ να λέει κάτι τέτοιο. Με πάρα πολύ. Είναι καθοριστική σημασία το πώς αξιολογείται ο κίνδυνος. Επαναλαμβάνω, ε, πρέπει να ισχύσει η αρχή της πρόληψης, ε, να υπάρξουν αυστηρότατοι περιορισμοί, αλλιώς να αποσυρθεί τον γλυκοσάτα από την αγορά. Η κυρία Ντορνάνο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Το ΙΑΡΚ λέει πως το γλυφοσάτ και τα παράγωγα που χρησιμοποιούνται με επικουρικές ουσίες οδηγούν σε κίνδυνο τοξικότητας. Αυτό αποτελεί επαρκή βάση για να θεωρήσουμε ότι τα προϊόντα που περιλαμβάνουν εγκλήφοζατ εξαιτίας των επικουρικών ουσιών ε, αποτελούν κίνδυνο για την υγεία. Από εκεί και περι λέει ότι πρέπει να καθορίσουμε την τοξικότητα του γλυφοζάτ και βασίζεται στο γεγονός ότι οι μελέτες για τα ζώα δεν έχουν ε, καταλήξει σε αποδείξεις για το αίτιο και το αιτιατό, ανάμεσα δηλαδή στη χρήση κλειφοζάτ και τον καρκίνο στον άνθρωπο. Δεν βρίσκω αρκετά σοβαρό το επιχείρημα αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, οι αποδείξεις τοξικότητας δεν πρέπει να περιμένουμε να αποδειχθούν πλήρως για να πάρουμε προληπτικά μέτρα. Και η Εύσυνη σαν να λέει ότι δεν υπάρχει κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Οπότε ρωτώ, τι γίνεται με την τοξικότητα για το περιβάλλον τότε, ε, για τη γη, για το έδαφο. Ζητήθηκε ευρία μελέτη για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε η κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εδώ όλοι δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στα συμπεράσματα της ΕΦΣΑ και του ΙΑΡΚ. Όντω οι μελέτε δεν έγιναν με τον ίδιο τρόπο, το ακούσαμε. Η μία είχε να κάνει με την ίδια τη χημική ουσία και η άλλη ε, χρησιμοποιεί και πρόσθετα στοιχεία, διαφορετικούς χημικούς τύπους δηλαδή. Η ΕΦΣΑ όμως είναι εκείνη που δίνει επιστημονικές συμβουλές στην Κομισιόν. Αν λοιπόν οι γνωμοδοτήσεις τη ΕΦΣΑ αμφισβητούνται, τότε τι την έχουμε την ΕΦΣΑ αν η Κομισιόν τελικά ε, δεν πρέπει να ακολουθεί τις νομοδοτήσεις της ΕΦΣΑ. Όπως καταλαβαίνετε έτσι χάνεται η αξιοπιστία. Αποδυναμώνεται η αξιοπιστία της ΕΦΣΑ. Κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε κάτι γι' αυτό. Τώρα δεύτερον πρέπει να βγούμε από το αδιέξοδο που βρισκόμαστε. Εγώ πιστεύω ότι η ΕΦΣΑ πρέπει να μπορεί να συνεχίσει τις δοκιμές για την ε, σύνδεση της δραστικής ουσίας με άλλα προσθετικά που χρησιμοποιούνται συνήθως. Και ένα από αυτά περιλαμβάνεται στο ριτς. Α, όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε περισσότερο πριν πάρουμε την τελική μας απόφαση για την άδεια ή την απαγόρευση του γλυφωσάτου. Ζητάω να τοποθετηθούμε βάσει επιστημονικών και λογικών δεδομένων. Ευχαριστούμε. Κυρία Πέλιερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούσαμε ήδη πολλά. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω για την παρουσίαση των μελετών. Σας ευχαριστώ που ήρθατε να συζητήσετε και μαζί μας. Δεν έχουμε προχωρήσει βέβαια καθόλου φοβάμαι. Θέλουμε τα επιστημονικά δεδομένα των ε, υπηρεσιών αυτών, αλλά μετά πρέπει να προχωρήσουμε εμείς στην πολιτική αξιολόγηση. Όταν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι καλά καταρτισμένοι χρησιμοποιούν αυτά τα προϊόντα, πρέπει να ξέρουν χρησιμοποιούμε πολύ το γλυφοζάτ. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και άλλα στοιχεία πέρα από την υγεία, την βιοπικιλότητα κτλ. Συνεπώς, εγώ θέλω να μάθω το εξή. Εσείς τι επιθυμείτε. Σας ζητάμε να αξιολογήσετε αυτό το προϊόν. Και θέλουμε από εσά αποτελέσματα. Είπατε ότι μπορεί να υπάρχουν νέα αποτελέσματα. Μπορείτε να μας πείτε τι το καινούριο ε, περιμένουμε που δεν είχαμε μέχρι τώρα στη διάθεσή μας. Θέλετε νέα εντολή να σας δώσουμε. Κύριε Εκάουτ, αν θέλετε τώρα το λόγο. Αν επιμένετε πρόεδρε, λέει ο κύριος Εκάουτ, ναι. Μια απλή ερώτηση έχω προς την Ιάρκα. Γιατί λίγο πολύ Αυτά που λέει σε εσά ο εκπρόσωπο ΕΦΣΑ είναι ότι η ΕΦΣΑ κάνει καλύτερα τη δουλειά τη από εσά. Εγώ έτσι συνοψίζω τόσα μα είπε η ΕΦΣΑ. Οπότε θα ήθελα να σα ακούσω να αντιδράτε σε αυτά που ακούσατε από την ΕΦΣΑ μετά τη δικιά σα παρουσίαση. Και προ την ΕΦΣΑ έχω δύο πλές ερωτήσει. Πρώτον, ισχυρίζεστε ότι έχετε χρησιμοποιήσει περισσότερε μελέτε. Πόσε από αυτέ τι μελέτε ε, μα έρχονται από τη βιομηχανία, από τον κλάδο. Πείτε μα ε, συγκεκριμένα. Δεύτερον, και αυτό ρωτήθηκε αρκετέ φορέ μέχρι τώρα, αλλά θέλω συγκεκριμένη απάντηση. Υπάρχει επιστολή προ την ΕΣΦΑ, προς την ΕΦΣΑ, η οποία επικρίνει τη διαφάνεια. Λέει ότι δεν ακολουθείτε τι διαδικασίε σωστά, ότι αφαιρείτε παραθέσει από τι μελέτε. Και εσεί εξακολουθείτε να ισχυρίζεστε ότι δουλεύετε με διαφάνεια. Λοιπόν, θέλω να ξέρω, ή οι 96 επιστήμονες ψεύδονται ή είσαστε υπερβολικά αισιόδοξοι όσον αφορά τη διαφάνεια της υπηρεσίας σας. Θέλω να μου απαντήσετε με σαφήνεια σε αυτό. Ευχαριστώ. Η κυρία Εύη. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ για τις δύο παρουσιάσεις, αλλά ήταν χρήσιμες μόνο στο ότι μου δημιουργήσαν περισσότερη σύγχυση. Θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ στους 96 εμπειρογνώμονες που νομίζω ότι προκαλούν ένα περαιτέρω στοιχείο σύγχυσης. Ε, μια άμεση ερώτηση. Η εμπορική παρουσίαση του προϊόντος της Μονσάντο είναι κάτι που χρησιμοποιείται στην πραγματικότητα, θα ήταν πιο σκόπιμο να έχουμε αξιολογήσεις ε, του τι χρησιμοποιούνται στην πραγματικότητα και όχι μόνο την ενεργό ουσία. Θα ζητήσω και από τις δύο, τα δύο υπηρεσίε τι χρησιμεύουν τα πρόσθετα τα οποία χρησιμοποιούνται στον αυτές νομίζω ότι για τη βελτίωση του προϊόντος, έτσι δεν είναι. Να αναφερθώ επίσης και στις μελέτες που ήδη μνημονεύτηκαν, οι εργασίες που δεν έχουν δημοσιευτεί και έχουν διαφορετική ε, σημασία με αυτές τις peer review. Όπως η ΕΦΣΑ αιτιολογεί, δικαιολογεί αυτήν την στάση της, και ως εκ του κάτι που είπαν και όλοι οι συνάδελφοι γιατί στην περίπτωση αυτή δεν χρησιμοποιείται ουσιαστικά και με τρόπο ε, σαφή και ξεκάθαρο η αρχή της ε, πρόληψης. Ευχαριστώ κύριε Ντόρφμαν. Ο κύριος Ντόρφμαν, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, δεν είναι σωστό για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως είναι η καρκινογέννηση να μην έχουμε χρόνο να τοποθετηθούμε. Βλέποντας όμως ε, το πώς παρουσιάζει το θέμα στον τύπο, έχω κάποιες αμφιβολίες. Αυτό το γλουφοσάτ συνδέεται με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και έχω κάποιες ε, αμφιβολίες. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι εδώ πρόκειται μόνο για τον γλουφοσάτ ή πρόκειται και γενικότερα για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Και βλέποντας κάποια παραδείγματα από το παρελθόν, ορισμένοι συνάδελφοι είπαν ότι η βιομηχανία θέλει να υπερασπιστεί αυτό το προϊόν. Βλέποντας όμως τις εναλλακτικέ λύσεις ε, και το κόστος αυτών των λύσεων που ε, αφορούν τους ίδιους τους παραγωγούς, η βιομηχανία πιθανόν ενδιαφέρεται να αποσυρθεί το γλυφοσάτ και να εμφανιστούν οι εναλλακτικέ λύσει. Ο συνάδελφο Χόισλε το είπε ότι ε, το γλυφοσάτ δεν είναι ένα τυχαίο προϊόν. Το γλυφοσάτ είναι το σημαντικότερο από τα φυτοφάρμακα. Δηλαδή δεν είναι ότι αν ε, το γλυκοσάτ αρχίσουμε να ξεχορτίζουμε με την τζουγκράνα. Ε, όσοι το πιστεύουν αυτό κάνουν λάθος. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα ήθελα να ερωτήσω αν εξαφανιστεί το γλυκοσάτ, τι θα γίνει με τις ε, υπόλοιπες εναλλακτικές λύσεις. Έχουν γίνει μελέτες για την τοξικότητα αυτών των εναλλακτικών λύσεων. Πραγματικά θα επιτύχουμε βελτίωση της κατάστασης αν αποσυρθεί το γλυκοσάρι. Ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας και τις επιδράσεις πάνω στις μέλισσες τέτοιων ουσιών. Ξέρουμε λοιπόν ότι είναι επικίνδυνο το γλυφοσάτο για καρκίνο. Εδώ λέει με σαφήνεια από την ΕΦΣΑ ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο, αλλά από την άλλη μεριά λέτε να υπάρχουν νέοι κανόνες όσον αφορά τη μελέτη της ουσίας αυτής για να δούμε τι υπόλοιπα μένουν στα τρόφιμα. Αν υπάρχει όμως τελικά ο κίνδυνος, γιατί εγώ έτσι καταλαβαίνω αυτό που λέτε, πόσο στα σοβαρά θα πάρουμε τις μελέτες που λένε ότι υπάρχει επικίνδυνοτητα. Τελικά πρόκειται για την υγεία του ανθρώπου. Ο κύριος Γιάρα. Εκτός μικροφώνου, δεν ακούγεται ο κύριος Γιάρ, δεν δουλεύει το μικρόφωνο του μάλλον. Kommt man links jetzt plötzlich. Also, oh, bei... <laughs> Ξαφνικά γίνομαι και εγώ πιο αριστερός, καθήμενος πιο αριστερά. Λοιπόν, η ΕΦΣΑ λέει ότι αν χρησιμοποιείτε σωστά το γλυκοσάτ ε, δεν υπάρχει πιθανότητα εμφάνιση καρκίνου. τι λέτε από αυτού. Και το δεύτερο ερώτημα είναι ότι τελικά ακόμα και αν χρησιμοποιούνται διάφορες ε, μάλλον οι ίδιες μέθοδοι καταλήγουμε σε διαφορετικό αποτέλεσμα. Τρίτο, εγώ ως ε, αδαής έχω την εντύπωση ότι η ΑΡΚ ε, δεν ταξινομεί ε, το προϊόν σε επικίνδυνη κατηγορία. Το βάζει σε δεύτερη κατηγορία όπως τα αστεροειδή. σε αυτήν την κατηγορία ανήκει και το κόκκινο κρέας, μα του ίδιου κινδύνου είναι το γλυκοσάτ. Ε, στην κατηγορία 1, ας πούμε, είναι ο καπνός που αφορά όσους καπνίζουν, ο αμύαντος, τα αλκοολικά ποτά, ε, το μεταποιημένο κρέας, όλα πάνε στην κατηγορία 1. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν είναι ότι από τη μια έχουμε μία μέθοδο, αλλά από την άλλη ε, δεν υπάρχει εμπειρία από την πρακτική εφαρμογή. Γιατί αλλιώς θα λέγαμε όποιος πίνει ένα ποτηράκι κρασί μια φορά τη βδομάδα θα πάθει καρκίνο. Ε, δεν γίνεται αυτό. Πρακτικά, τι έχετε να μας προτείνετε όσον αφορά αυτά τα αποτελέσματα. Η κυρία Ρής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χάος επικρατεί εδώ και χρόνια μελετών ε, έχει συμβουλευτεί με εκατοντάδες εμπειρογνώμονες η ΕΦΣΑ και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κάποια κατάληξη αλλά εγώ μια περίπτωση όπως σημερινή πρώτη φορά την αντιμετωπίζω ζητάμε δηλαδή, την Κομισιόν και σε εμά να λάβουμε μια απόφαση. Βρισκόμαστε σε αδίέξοδο νομίζω όπως το είπε η κυρία Γκροστέτ συμφωνώ με πολλά από τα επιχειρήματα που ακούστηκαν ε, κατά τη διάρκεια τη συζήτηση ε, παρατηρώ ότι οι παρεμβάσει τη κυρία Γκροστέτ και τη Διαβάση βρίσκονταν στο γενικό σχήματο, κάτι το σπάνιο και διερωτώ με ε, εδώ έχουμε κάποια ευκαιρία αν ξέρουμε λοιπόν ποια είναι η ενεργοσυδία και όχι τα πρόσθετα τα οποία παρουσιάζουν πρόβλημα οι διαφορετικές διαδικασίες οι οποίες εφαρμόζονται και μάλλον εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια της εξέτασης των προβλήματος και των μελετών. Αντί λοιπόν να πρέπει να δώσουμε ένα τέλος εδώ θα πρέπει να συνεχίσουμε να αναζητάμε τις αποδείξεις διότι περί αποδείξεων πρόκειται. Αυτές ζητάμε, ζητάμε, ακούμε για την αρχή της απαγόρευσης ή για της πρόληψης. Ναι, είναι μια απόφαση κάπως συγκινησιακή και, κάπως και μάλλον εύκολη και ο Ντόρφμαν με κάλυψε, αλλά δεν ήταν σημερινά το σημερινό ζήτημα, αλλά ποιες είναι οι εναλλακτικέ λύσεις. Ένας άλλος Γερμανός συνάδελφος μίλησε για μια μείωση κατά 40% των ε, συγκομιδών που γίνονται με το Roundup. Και τι γίνεται. Εγώ θα ήθελα να ακούσω όσες περισσότερες αντιδράσεις ε, υπάρχουν, αλλά είμαι της άποψης ότι το καλύτερο δεν είναι εχθρός του καλού. Πάντως από τη σημερινή συζήτηση δεν έχει προκύψει τίποτα. Ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση και τώρα αναμένουμε τις απαντήσεις. Έχουμε διερμηνία για 10 λεπτά ακόμα, μετά θα συνεχίσουμε στα αγγλικά, λυπάμαι. Ήταν ε, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, δίνω το λόγο λοιπόν στην ERC και μετά στην ΕΦΣΑ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ε, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και τις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ορισμένα θέματα που απευθύνθηκαν ε, στον οργανισμό μας. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι αν τελειώσουμε τη συζήτηση καταλήγοντας ε, στο ότι δεν ήταν ικανοποιητικό το αποτέλεσμα της συζήτησης, αυτό δεν θα ήταν σωστό. Εγώ δεν μ' αρέσει να πούμε είτε ισχύει το ένα είτε ισχύει το άλλο. Κατά τα άλλα, να σας πω επίσης ότι αυτή η αξιολόγηση δεν ήταν περίπλοκη για τον οργανισμό μας. Εμείς ε, χρησιμοποίησαμε τη στάνταρτ μέθοδό μας ε, που είναι ευρέως αποδεκτή τα τελευταία 40 χρόνια. Για να απαντήσω σε μία από τις ερωτήσεις. Κοιτάξτε, η δική μας η ταξινόμηση μας οδήγησε στο ότι η συγκεκριμένη αυτή ουσία μπορεί πράγματι να προκαλέσει καρκίνο. Ε, και υπάρχουν και άλλες ουσίες σε αυτή την κατηγορία. Να πω μερικά πράγματα για να ξεκαθαρίσω τη συζήτηση. Πρώτα απ' όλα, να είμαι απόλυτα σαφή ότι ο δικός μας οργανισμός δεν περιορίζει την ανάλυση ε, σε ε, διάφορες ε, τοποθετήσεις ε, για την καρκινογέννηση, η πιθανότητα καρκινογέννησης σε ζώα ή για την πρόκληση ζημιάς στο DNA. Πιστεύω λοιπόν ότι ίσως υπάρχει εδώ κάποια παρεξήγηση σχετικά με την επιστημονική βάση. Επίσης, ε, τα δεδομένα, ε, πιθανότητα εμφάνισης καρκινογέννησης στα ζώα, ε, αυτά ισχύουν και γενικότερα σχετικά με τοξικότητα. Τώρα, ως πρώτα τεστ, τα χρησιμοποιούμε για να διαπιστώσουμε μία τάση την τάση που διαφαίνεται. Αυτή είναι μία στάνταρ μέθοδος που χρησιμοποιείται για να αναλύσουμε τα τεστ καρκινογέννησης στα ζώα. Δεν χρησιμοποιούμε εδώ τίποτα το περίεργο. Η τοξικότητα στα γονίδια, στα κύτταρα, έγιναν μετρήσεις πριν και μετά την έκθεση σε πραγματικά επίπεδα ε, χρησιμοποίησης ε, με ράντισμα του ε, γλυκοσάτ. Οι επιδημιολογικές μελέτες εξετάζουν ότι πραγματικά χρησιμοποιείται στον κόσμο συγκεκριμένες ενώσεις, αλλά πρέπει να επισημάνουμε ότι οι ενώσεις αυτές διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική τους χρήση, διαφέρουν γεωγραφικά και με άλλα κριτήρια στις διάφορες υπήρους κοινό βέβαια παράγων ίσως να είναι το γλυκοσάτ. Και κάτι άλλο που θέλω να πω. Προκλήθηκε η εντύπωση ότι ο δικός μας οργανισμός ε, δεν προέβη σε εκτεταμένες μελέτες, ότι δεν κάναμε συγκρίσεις ε, με διάφορα άλλα στοιχεία που χρησιμοποιεί η ΕΦΣΑ. Δεν πρόκειται για την ποιότητα, μάλλον για την ποσότητα, αλλά για την ποιότητα των πληροφοριών. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ενδελεχής ε, έλεγχος να κοινοποιηθούν τα στοιχεία και άλλοι να κρίνουν ε, τα στοιχεία αυτά κατά πόσο οδηγούν στην ε, καρκινογέννηση ή όχι. Είναι λοιπόν αλήθεια ότι εξετάσαμε λιγότερες πληροφορίες και δεν λάβαμε υπόψη μας ε, μελέτες που δεν έχουν κοινοποιηθεί. Ο εντελεχής έλεγχος είναι πολύ σημαντικός όσον αφορά την επιστημονική μέθοδο πρέπει κανείς να μπορεί να ακούει ε, και βεβαίως και να εξετάζει και άλλες μελέτες. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία που θα ήθελα να φέρω ε, προς διευκρίνηση, κυρίως όσον αφορά τις ε, ενώσεις και τα δεδομένα που χρησιμοποίησαμε. Αν είχαμε περισσότερες πληροφορίες για την καρκινογέννηση ή για την κυταροτοξικότητα, ε, αυτά δεν θα άλλαζαν την αξιολόγησή μας γιατί ε, ήταν θετικέ οι μελέτες τόσο ε, στα κύτταρα των ζώων όσο και των ανθρώπων. Αυτό ήταν απόλυτα σαφές για την ομάδα εργασίας μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε και τώρα η ΕΦΣΑ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Χωσέ για μια σύντομη επιστημονική μελέτη και εγώ θα κάνω την ανακεφαλαίωση. Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ για όλα τα σχόλια. Η αξιολόγηση της ΕΦΣΑ γίνεται για τη δραστική ουσία γιατί έτσι λέει ο κανονισμός. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει η έγκριση της δραστικής ουσίας και υπάρχει μια peer review που γίνεται από την ΕΦΣΑ και μετά είναι ευθύνη των χωρών μελών να κάνουν την αξιολόγηση και να αποφασίσουν για την άδεια ή όχι κάθε προϊόντος που μπορεί σε διαφορετική σύνθεση να χρησιμοποιούν τις ουσίες που έχουν εγκρίνει οι χώρες μέλη. Όσον αφορά τώρα την τοξικότητα και την επικινδυνότητα καρκινογένεσης, οι γνώσεις μας είναι διαφορετικές. Μπορείτε να πάτε στις κατευθυντήριες γραμμές ε, του site της υπηρεσίας ε, για τις χημικές ουσίες η αξιολόγηση γίνεται μόνο ο, για δύο δηλαδή συνδυασμένες ουσίες την κάνετε την αξιολόγηση μόνο όταν υπάρχουν ενδείξεις για επικινδυνότητα καρκινογέννησης. Και μετά κατά πόσο κατά πόσο είναι από μόνα τους η σύνθεση των ουσιών η οποία οδηγεί στην επικινδυνότητα. Έχουμε λάβει υπόψη μας όλες τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες και συστήνουμε στις χώρες μέλη να ελέγξουν για την ε, τοξικότητα όλα τα συθετικά. Οι χώρες μέλη έχουν ε, ένα ντοσιέ όπου εντοπίζονται όλα τα συνθετικά. Για τις μελέτες πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλες τις πληροφορίες που έχουν χρησιμοποιηθεί για κάθε ουσία, όχι μόνο για το γλύφασατ μόνο του, αλλά και για όλα τα συστατικά, τον βαθμό καθαρότητας, για να δούμε τι είναι αυτό που οδηγεί ή όχι σε τοξικότητα. Και το κάνουμε αυτό και για τον κλειφασέτο όσον αφορά την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Αν πούμε ότι δεν έχει να κάνει το αποτέλεσμα με τη δραστική ουσία αλλά με ένα άλλο συνθετικό, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτό μπορεί να ισχύει και για άλλες ε, τότε χημικές ενώσεις. Γιατί κάποιες ε, συνθετικές ουσίες είναι τοξικές και κάποιες όχι που έχουν την ίδια δραστική ουσία. Τα συμπεράσματα δημοσιεύτηκαν αλλά δεν έχουμε αρκετέ πληροφορίε για να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει η τοξικότητα αυτή. Όσον αφορά την ε, διαφάνεια της μεθοδολογίας και τι πληροφορίε που είναι δημοσιευμένες ή όχι. Όλες οι πληροφορίες όσον αφορά την αξιολόγηση τη ΕΦΣΑ είναι δημόσιες. Ο κανονισμός 1107 μας το επιβάλλει. Κάθε μελέτη από τις 24 εταιρείε που έδωσαν μελέτες δημοσιεύτηκαν από την αρχή και υπάρχει και δημόσια διαβούλευση. Είναι σημαντικό να πούμε επίσης ότι όσον αφορά την επικεντρινότητα καρκινογένεσης, η ΕΦΣΑ χρησιμοποιεί μελέτες, λέτε, από την βιομηχανία. Μία ήταν και είχαμε πει ότι δεν ισχύει για την αξιολόγηση. Χρησιμοποιούμε λοιπόν πληροφορίες. Είχαν γίνει και άλλες μελέτες νωρίτερα. Η ΕΦΣΑ πάντως έχει το ίδιο επίπεδο πληροφορίας και για άλλες μελέτες και για τις μελέτες της ΕΦΣΑ. Όσον αφορά τη τοξικότητα της δραστικής ουσίας, δεν κάνουμε συγκρίσεις βέβαια, αλλά κάπου 40-50 διαφορετικές δραστικές ουσίες αναλύουμε. Και τα αποτελέσματα μας δεν έχουν να κάνουν μόνο με την επικίνδυνοτητα καρκινογένεσης, αλλά και με άλλες ε, μελέτες και